Παρακαλώ, ξεκινάμε την Επιτροπή μας και πάλι σήμερα το απόγευμα στις θέσεις σας όλοι. Innanzitutto voglio salutare e ringraziare della loro presenza θα ήθελα να ευχαριστήσουμε την παρουσία τους μια ομάδα επισκεπτών από τον κύριο Ταραμπέλα, ε, που είναι γεωργοί και είναι και γεωπόνοι και τους ευχαριστούμε όλους που ήρθαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε λοιπόν τους επισκέπτες μας για την παρουσία τους εδώ, για την παρουσία τους. Να ξεκινήσουμε. Για να μπούμε στο ψαχνό. Ε, ορίζοντας του 2020 για την ΚΑΠ λοιπόν, ε, το σημαντικότερο θέμα είναι αναθεώρηση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ε, το 18 Νοεμβρίου έκανε παρουσίαση ο Επίτροπος και έτσι μπήκαμε στο κυρίως θέμα και τους ε, επόμενους μήνες κάθε μέρα θα μας απασχολεί αυτό το θέμα για να δούμε πώς θα χαράξουμε μια φιλόδοξη κάποια το μέλλον ε, που να αποκνίζει τις καθημερινές προκλήσεις ε, και να έχει μια προοπτική για να συνδυάσει τις υπηρεσίες, ε, τα αγαθά και με τις αναγκαίες εγγυήσει για υποστήριξη οικονομικής του Γιώργους. Και αρκετές φορές τώρα την τελευταία χρονιά το παρατηρήσαμε ότι η θέση ισχύ της συνθήκης της Σαββόνας μας έδωσε περισσότερες ευθύνες, μας φόρτωσε περισσότερες ευθύνες σε σχέση με το παρελθόν και έχουμε πρωταγωνιστικό πια ρόλο θεσμικά και μπορούμε να επηρεάσουμε ιδιαίτερα τα πράγματα στις διαδικασίες έγκρισης και επαφής και να δούμε τα άσχημα σημεία πώς θα τα διαγράψουμε, πώς θα τα βαλείψουμε και αυτά στα πλαίσια των Αρκαιώσεων της Επιτροπής. Έχετε στα αγγλικά το κείμενο, το έγγραφα αυτό και σε μία εβδομάδα θα το έχετε και σε όλες τις υπόλοιπες γλώσσες. Μια παρόμοια περίληψη όμως υπάρχει έτσι κι αλλιώς στις ε, Θα ήθελα να χαιρετήσω τον κύριο Τάσο Ανιώτη από την Επιτροπή, από την Γενική Διάθεση Γεωργίας. Σε ευχαριστούμε Τάσο που είσαι εδώ ανάμεσά μας και θα μας βοηθήσεις για περισσότερες λεπτομέρειες για να απαντήσουμε σε όλα αυτά που μας απασχολούν. Θα ήθελα να δώσω το λόγο αμέσως στον Άλμπερντες ο οποίος θα μας κάνει μια εισαγωγή στο θέμα μας σήμερα το απόγευμα. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους και επίσης από την ε, Ιταλική Συνομοσπονδία Αγροτών θα ήθελα να του ευχαριστήσω για την παρουσία τους εδώ στην Επιτροπή μας σήμερα το απόγευμα. Αλμπερντές, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, Αγαπητοί διοργανωτές της σημερινής συνεδρίασης και μέλη της Επιτροπής, θα αναφερθώ σύντομα στο περιεχόμενο της ε, έκθεσης. Ευχαριστώ και την ομάδα εργασίας που ήδη έχει θέσει μια σειρά ερωτημάτων και μετά από την υποβολή της έκθεσης αυτής είπα ότι αποτελεί μια πολύ καλή βάση συζήτησης αλλά δίνει το έναυσμα και για περαιτέρω συζητήσεις. 74 ερωτήματα ή ζητήματα θίγει η ομάδα εργασίας 74 τα οποία θα πρέπει τους ερχόμενους μήνες να απαντηθούν από την Κομισιόν. Η πρόταση της Κομισιόν παραμένει ανοιχτή σε πολλά θέματα ακόμα, οπότε έχουμε μια θαυμάσια ευκαιρία στο Κοινοβούλιο να διαμορφώσουμε την έκθεσή μας ε, ακόμα πιο περιεκτικά για να τη συζητήσουμε στην Επιτροπή Γεωργίας, έτσι ώστε η Επιτροπή μας εδώ να παρουσιάσει μια ισχυρή έκθεση. Ελπίζω ε, να παραμείνει η δέσμευση στους δύο πυλώνες παρόλο που έχουμε ακόμα τόσα θέματα να συζητήσουμε και ελπίζω ε, να χρηματοδοτηθεί στο 100% ο πρώτος πυλώνας. Αυτό είναι αναμφισβήτητο το ότι χρειάζεται και συγχρηματοδότηση στο δεύτερο πυλώνα. Σημερίζουμε την άποψη της Κομισιόν ότι οι άμεσες πληρωμές μετά το 2013 θα πρέπει να κατανεμηθούν πιο θεμητά, πιο δίκαια μεταξύ των κρατών μελών και δεν μπορούν να παραμείνουν για ορισμένα κράτη-μέλη στο σημερινό ύψος. Όμως θα πρέπει να σκεφτούμε όλοι, όπως το έχουμε συζητήσει στην Επιτροπή, ότι οι αριθμοί τους οποίους συζητάμε σήμερα μεταξύ νέων και παλαιότερων κρατών θα αλλάξουν μέχρι το 2013. Τα στοιχεία αυτά θα αλλάξουν. Στα παλαιά κράτη-μέλη η αφετηρία μας ήταν το 2008, η βάση μας. Και είχαμε κατά μέσο όρο 288 ευρώ κατά εκτάρια το, το 2008 και στα νέα κράτη-μέλη είχαμε μόνο 98 ευρώ. Όμως μέχρι το 2013 αυτό θα αλλάξει διότι στα παλιά κρατημέλη παραμένει το παλαιό ποσό 2,88 ενώ στα νέα ε, αυξάνεται σε 192. Η διαφορά δηλαδή μεταξύ παλαιότερων και νέων είναι περίπου, θα είναι περίπου 100 ευρώ. Οπότε οι επιπτώσεις δεν είναι τόσο δραματικές όπως πολλές φορές παρουσιάζονται. Δεδομένου ότι δύο είναι ο μέσος όρος της έκτασης των παλαιότερων έναντι των νέων κρατών μελών. Οπότε, η ύψωση αυτή του ποσού των άμεσων πληρωμών επαρκεί για να κατανοηθούν πιο δίκαια οι πληρωμές αυτές. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι μετά το 2014 χρειαζόμαστε μεταβατικές περιόδους. Οι περισσότερες επιφυλάξεις μου επικεντρώνονται στον πρώτο πυλώνα με τις προτάσεις της Κομισιόν. Σίγουρα θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και εδώ στην Επιτροπή αλλά και από τον κλάδο, από τους ενδιαφερόμενους και τις διάφορες διοργικές ενώσεις και συλλόγους έχω ακούσει πολλές αντιρρήσεις μετά την παρουσίαση της ανακοίνωσης της Κομισιόν πλην ενός κανένας δεν μου είπε ότι η πρόταση αυτή της Κομισιόν είναι πρακτικά εφαρμόσιμη. Όλοι έχουν μεγάλες ανησυχίες ότι εάν εφαρμοστεί τέτοια πρόταση της Κομισιόν θα έχουμε μια τεράστια επιπλέον επιβάρυνση της γραφειοκρατίας. Επίσης αυτό που πολλές φορές αναφέρεται είναι ότι πρέπει να δικαιολογήσουμε στην κοινή γνώμη γιατί έχουμε τις αντιστασμιστικές πληρωμές στον αγροτικό τομέα. Και πώς δικαιολογούμε την πολιτική του πρώτου πυλώνα. Είναι λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, πολύ σοβαρή η διάθεση, το ύψος των κονδυλίων που διαθέτουμε. Εάν εκα, θέλαμε ένα budget με 150 ευρώ στον πρώτο πυλώνα, δεν θα χρειαζόταν μεγάλα έξοδα στον πράσινο τομέα. Εάν όμως θέλουμε 272 ευρώ, τότε θα αλλάζει η κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν ε, να λάβουμε υπόψη μας για να έχει νομοθετικό περιεχόμενο βεβαίως, νομοθετική βάση η έξεση, ποια κονδύλια ακριβώς είναι διαθέσιμα. Εάν είναι κάποιος εκπρόσωπος του τύπου εδώ, τα πράγματα θα διαρρεύσουν στην δημοσιότητα. Οι γεωργικές ε, δαπάνες στην ε, Ευρώπη αναφέρονται συνέχεια στον τύπο ε, και μέχρι το 2000 η αγροτική πολιτική επικρινόταν συνέχεια. Έπρεπε λοιπόν συνέχεια να δικαιολογήσουμε την πολιτική μας ε, στη δεκαετία του 70 είχαμε 87% του κόστους του ευρωπαϊκού μπάτζετ ήταν στο γεωργικό τομέα, καλύπτεται από τον αγροτικό τομέα τη δεκαετία του 70. Εν συνεχεία το ποσοστό αυτό ήταν πάντοτε πολύ υψηλό. Πρέπει λοιπόν τώρα να βρούμε ένα συμβιβασμό ώστε να υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ του πρώτου και δεύτερου πυλώνα, να λάβουμε υπόψη περισσότερο τον πράσινο παράγοντα στον δεύτερο πυλώνα και να βρούμε καλύτερους και ακριβέστερους ορισμούς. Όταν ε, μιλάμε για ανώτατα κατόφλια, πρέπει ανώτατα όρια, πρέπει να σκεφτούμε πώς θα διαμορφώσουμε αυτά τα κριτήρια, αυτά τα οριακά στοιχεία, διότι οι παραγωγοί έχουν πολλές διαφορετικές απόψεις ε, πρέπει να βρούμε σαφείς ορισμούς για το πού σταματάνε τα, τα μέτρα μας, ποια είναι τα όρια, ποια είναι η οριακή γραμμή ή το οριακό στοιχείο. Ε, η άποψη της Κομισιόν ότι στις άμεσες πληρωμές θα πρέπει να εφαρμοστεί το περιφερειακό μοντέλο και ότι θα πρέπει να εφαρμόσει την ίδια πολιτική στις άμεσες πληρωμές όπως και στα περιφερειακά κονδύλια, στην περιφερειακή πολιτική. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε ίση μεταχείριση για τις μικρές μονάδες. Έχουμε 13,5 παραγωγούς με τις σημερινές στατιστικές. Εάν θέλουμε να εισαγάγουμε επιπλέον πριν, θα θα φύγουν τα 13, θα χάσουμε 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνω λοιπόν, εάν θέλουμε επιπλέον δαπάνες για τους μικροπαραγωγούς, πρέπει να βρούμε ένα σωστό ορισμό των ο, ε, ανωτάτων ε, οροφών για να είναι δίκαιες ε, οι πληρωμές μας. Ε, ε, ε, παρέμβαση και ποια, μέσα της παρέμβασης θα διατηρήσουμε πια αυτές τις συζητήσεις τις έχουμε ήδη κάνει στην Επιτροπή μας και οι συζητήσεις οι ενδοπολιτικές με τις ομάδες δηλαδή οι συζητήσεις που έχω κάνει δείχνουν ότι θα παραμείνουν οι μηχανισμοί που ισχύουν εάν καταργήσουμε τους μηχανισμούς και συνεχεία διαπιστώσουμε λόγω διακοιμάσεων των αγορών ότι πρέπει να επαναφέρουμε τους μηχανισμούς δεν θα μπορέσουμε να το πράξουμε αυτό πολύ γρήγορα για να παρέμβουμε. Σύμφωνο στην ανακοίνωση της Κομισιόν ότι τα αντισταθμιστικά ποσά για τις απομακρυσμένες και εξαιρετικά απομακρυσμένες περιοχές πρέπει να παραμείνουν στο δεύτερο πυλώνα και ότι θα πρέπει να υπάρχουν προαιρετικά μέτρα όχι υποχρεωτικά τα οποία θα καλύπτονται από το ελάχιστο επίπεδο συγχρηματοδότησης μέχρι 10%. Και ότι για μέτρα τα οποία έχουν υψηλότερη προτεραιότητα μπορούμε να ε, εφαρμόσουμε υψηλότερο βαθμό συγχρηματοδότησης. Η συγχρηματοδότηση θα βασίζεται βασικά στην χαμηλότερη δυνατή παρέμβαση των δημοσίων πιστώσεων. Πρέπει λοιπόν να οριοθετήσουμε ε, την διαμόρφωση του δεύτερου πυλώνα για να έχουμε και μια ξεκάθαρη διαρθρωτική πολιτική. Πρέπει να ενισχύσουμε και την, τον τομέα της έρευνας μέσα στην έκθεση για να μην ε, παραμείνουμε ουραγοί στην Ευρώπη και η έρευνα λοιπόν πρέπει να αναφερθεί στην έκθεση και να βρούμε έναν θεμητό συμβιβασμό πέραν των ε, πολιτικών ενδιαφερόντων των διαφόρων ομάδων έχουμε συνεργαστεί και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε καλά με τον αρμόδιο επίτροφο. Αυτά είχα, είχα να παρατηρήσω εισαγωγικά και ε, δυστυχώς επειδή έχουμε ένα πένθος στην οικογένεια πρέπει να φύγω σε μία ώρα και σας ζητώ την κατανόησή σας. Δυστυχώς πρέπει να γυρίσω στην πατρίδα μου. Σας ευχαριστώ για αυτήν την ευκαιρία που μου δώσετε για την πρώτη σύντομη παρέμβαση στο θέμα. Πολύ καλά, σε ευχαριστούμε. Έχουμε πολύ υλικό στα χέρια μας τώρα πια. Ξεκινάμε τη συζήτηση και θα δώσουμε το λόγο στον Στεφάν Λεφόλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μας έκανε μια γενική παρουσίαση ο Αλμπέρ της δικής του προσέγγισης. Θα πρέπει να το συζητήσουμε και πάλι μαζί θα την παρακολουθήσω από πλευρά σοσιαλιστών αυτή την έκθεση. Θέλω να σας πω το εξής. Έχουμε εκατοντάδες σημεία στα οποία θα ήθελα να επιμείνω. Την οργάνωση ανάμεσα στους δύο πυλώνες. Για να δούμε πιο ξεκάθαρα τα πράγματα αυτά που πρότεινε ο Επίτροπο. πάει προς τη μία κατεύθυνση και ο πρώτος πυλώνα να έχουμε μια εναρμόνιση εκεί όλων των ενισχύσεων. Και ο δεύτερος πυλώνα που να πηγαίνει στις ενισχύσει εκείνε που αφορούν πολιετή περιόδους. Είναι σημαντικά αυτά τα πράγματα, πρέπει να τα δούμε, να τα εξετάσουμε, να τα συζητήσουμε από κοινού για να δούμε από τεχνική πλευρά πώ θα μπορέσουμε να ε, προσαρμοστούμε. Εντάξει, ένα μέρος από αυτέ τις δημιουργικές ενισχύσεις του πρώτου πυλώνα θα μπορούσαν να ενισχύσουν αυτό το θέμα που τίθεται, δηλαδή τη διατήρηση της γεωργικής δραστηριότητας σε περιοχές που δεν είναι και τόσο εύκολες, εκείνες που έχουν μειονεκτήματα ενδεχόμενα. Το δεύτερο σημείο, το είπε έχει να κάνει με το θέμα, πώς να σας το πω τώρα, κοινωνική απασχόληση. Τι εννοώ τις μικρές εκμεταλλεύσεις. μα είπε ορισμένου αριθμούς, θα πρέπει να τα εξετάσουμε αυτά, να δούμε τι θα μπορέσει να γίνει στον τομέα αυτό. Αλλά σημαντικό θα είναι κατά την απόψή μα να τα δούμε αυτά τα πράγματα, να δούμε την ανάγκη που υπάρχει, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για τις μικρές εκμεταλλεύσει για να απλωστευθεί κάπω η διαχειριστική τη πολιτική πολιτικής και έτσι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα καθεστώ ε, πραγματικά για όλες αυτές τις μικρές εκμεταλλεύσει, ε, τον απασχολεί τον Επίτροπο και εμείς προ αυτήν την κατεύθυνση θα πρέπει να τον βοηθήσουμε. Τώρα, στο σύνολο αυτό για την κοινωνική απασχόληση, άλλο ένα στοιχείο πολύ σημαντικό για μένα είναι ανάμεσα στι ενισχύσει και στον ενεργό πληθυσμό τον αγροτικό που λέει και ο Επίτροπο. Και πάνω σε αυτό θα πρέπει η Επίτροπη Γεωργία προ αυτήν την κατεύθυνση πραγματικά να εργαστεί και να δώσουμε ενισχύσει ε, χωρί να έχουμε μια παραγωγή από την άλλη μεριά ή ούτε γεωργοί καθόλου να μην υπάρχουν. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι έχει με ιδιαίτερη σημασία και η Επιτροπή Γεωργία θα πρέπει να υποστηρίξει αυτήν την κατεύθυνση, δηλαδή πίσω από αυτή τη ενισχύσει δημόσια θα πρέπει να υπάρξει και απασχόληση γεωργική και να μην δίνουμε ενισχύσει, να μην προσφέρουμε ενισχύσει μόνο και μόνο για να δίνουμε χρήματα και εισόδημα στου γεωργού. Ε, εντάξει, οτιδήποτε ε, ακούγεται έτσι σαν να έχει ιδιαίτερη σημασία. Και ακόμα κάτι για την ΚΑΠ, αυτό το ε, ναι, οικολογική μετάβαση που θα πρέπει να γίνει σε αυτή την κοινή γεωργική πολιτική και στην γεωργία την ευρωπαϊκή και ο στόχος, και εντάξει όλοι μαζί το ξέρουμε εδώ, είναι σαφές εδώ στην Επιτροπή Γεωργίας, θα πρέπει να είναι κανείς οικονομικά αποδοτικός και οικολογικά αποδοτικός. Δεν μπορεί το ένα αντίθετο στο άλλο. Και εδώ με τη συζήτηση με τον Αλμπέρ εδώ πάνω σε αυτό και για το κλίμα επίση. Έστω και αν χαμηλώνει η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχουν ορισμένα θέματα στα, ε, στα ε, περί κλίματο που είναι αντίθετα, είναι εμπόδιο. Λοιπόν, θα πρέπει να το δούμε και στην πρόταση του Επιτρόπου για να μπορέσουμε να ε, προσαρμόσουμε καλύτερα του δικού μα στόχου. Αυτό που θα μπορεί να γίνει από την Επιτροπή. Πώς το αποκαλέσω τώρα, είναι κάπως ε, συμβατικό αυτό εναλλακτική ε, με, με, καλλιέργεια η μία μετά την άλλη και λοιπά, όλα αυτά δεν ξέρω, αλλά υπάρχουν ε, έτσι κι ήδη αυτή η οικοποθετικότητα συμμόρφωση ανάλογα και πρότυπα που θα μπορέσουν να μας επιτρέψουν αυτή την απόδοση και την οικολογική και την αγροτική. Αυτό είναι για μένα το τρίτο σημείο, ιδιαίτερα σημαντικό, Αλμπέρ. Πάνω σε αυτό η Επιτροπή Γεωργίας θα πρέπει να εργαστεί και μάλιστα με ιδιαίτερο και συγκεκριμένο τρόπο. Έχουμε ιδιαίτερου προσανατολισμού. Ε, πάνω σε αυτό είναι πολύ σημαντικό και το δεύτερο ε, πυλώνα εδώ η πολιτική για το περιβάλλον. Και όλα αυτά μπορούν να γίνει. Αυτέ οι συμφωνίε όπω με τον Ζον Ντάιεν με την έκθεσή του θα πρέπει και εκεί να μπορέσουμε να είμαστε ακριβέστεροι και θα πρέπει ταυτόχρονα να να επιτελέσουμε μια εργασία ανάλυση έρευνα πάνω σε αυτό το τομέα. Τελευταίο σημείο που είπε επίση και έδειξε ο Άλμπερ είναι οτιδήποτε έχει να σχέση με τη ρύθμιση των αγορών. Για να δούμε. Εδώ λοιπόν να προσπαθήσουμε όσο γίνεται να ελέγξουμε στα μέτρα του δυνατού τα δύο εξή φαινόμενα. Το πρώτο φαινόμενο, αυτό της κρίσης, χρειάζεται μια δημόσια επέμβαση παρότι ότι ίσως υπάρχουν και ορισμένα συστήματα εξασφάλισης, το πούμε έτσι. Αλλά όταν είναι βαθιά η κρίση, πολύ βαθιά, ξέρουμε ότι μια κάποια στιγμή είτε μια, μια ασθένεια για τα ζώα ή το, άλλο, πολύ βαθιές κρίσεις θα πρέπει ακριβώς επιζωτής, θα πρέπει να τα λύνουμε αυτά τα προβλήματα και να επεμβαίνουμε. Και τα είδαμε αρκετά, είδαμε αρκετές και είδαμε ότι αυτά τα πράγματα βαραίνουν ιδιαίτερα. Το δεύτερο θέμα τώρα ε, για σιγά ρύθμιση είναι ότι οι τιμές κυμαίνονται από εδώ και από εκεί. Τι γίνεται, να αποφύγουμε οι τιμέ από το 120 ας πούμε σε 130 σαν δίκτυ να πάνε αλλού στο 60-70 μια κάποια στιγμή, δηλαδή μια κάποια χρονική στιγμή αργότερα. Αυτό το θέμα τίθεται και σαν ερώτημα και θα πρέπει πρώτο σημείο να διατηρηθεί ο μηχανισμό παρέμβαση σημερινό. Δεν μπορούμε να δεχτούμε έτσι να καταργηθεί κάτι, έστω και αν είναι με μηδενικό ποσοστό. Εντάξει, συμφωνώ κοίταμε με την κρίση των γαλακτοκομικών του Γαλακτό, αν είχε καταργηθεί κάθε μηχανικό παρέμβαση σε αυτόν τον απολογισμό τη. Α ε, την πούμε έτσι, υγεία. Όταν ήρθε η κρίση τότε ε, δεν θα είχαμε κανένα εργαλείο στη διάθεσή μα για να μπορέσουμε να παρέμβουμε. Λοιπόν αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί. Και θα πρέπει να διατηρηθεί, εντάξει ισχύει αυτό. Και ταυτόχρονα θα πρέπει να το συλλογιστούμε για να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε καλύτερα ακόμα να ρυθμίσουμε τα πράγματα και να αποφύγουμε έτσι να διακυμαίνονται τόσο οι τιμέ. Είναι το τέταρτο σημείο που κατά την απόψη μου είναι σημαντικό. Εδώ λοιπόν το επόμενο σημείο, με αυτά τα τέσσερα σημεία, τα κύρια σημεία τη όλη συζήτηση, θα πρέπει ε, σαν στόχο να διατηρήσουμε αυτό που λέει ο Ζωσντάιερ και τι σημαίνει. Το ότι δεν θα δεχτούμε μια επανεθνικοποίηση της κοινή γεωργικής πολιτικής μέσω οποιοδήποτε ε, τρόπου τεχνάσματος κλπ. Και δεύτερο, να περιορίσουμε αυτή τη συγχρηματοδότηση στο ε, Όπω έχει σήμερα η κατάσταση. Ναι, ναι, αυτές ήταν υποχρεώσει του Ευρωκοινοβουλίου που είχε αναλάβει, πολύ σημαντικέ και θα πρόβλημα μια συζήτηση για τις ε, δημοσιονομικές προοπτικές, επανοργάνωση του γενικού προϋπολογισμού ε, αυτό και τη γεωργίας θα προταθεί και θα πρέπει να δούμε την συνδυασμό ανάμεσα στην εξασφάλιση επιτόπου και στον γεωργικό προβλεσμό. Πάνω σε αυτά θα πρέπει να πρέσουμε ιδιαίτερα αυτά και μετά από την παρέμβαση του Άμπλμπερ. Αυτά είναι τα πέντε σημεία τα οποία κατά την απόψή μου πρέπει να προσέξουμε με πρωτοβουλίες, ε, συζητήσεις, ώστε η Επιτροπή Γεωργίας, όπως τότε στην έκθεση του Ζορντάιν, να μπορέσουμε να δείξουμε τη συνοχή μας όσο γίνεται περισσότερο, με ισχυρή θέση για να βαρύνουμε, να περάσουμε τις αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν ρυθμιστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πολύ καλά. Σε ευχαριστούμε, Στεφάν. Τώρα, ο Μάρκ Ταραμπέλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο Στεφάν Λεφόλ είπε τα κύρια που έπρεπε να υποθούν ε, σχετικά με τον Λεμπέρ. Ναι, πρόκειται για μια άριστη βάση εργασία στο έγγραφο αυτό τη Επιτροπή, αλλά παραμένουν πολλά θέματα ανοιχτά. Τώρα εντάξει, και αν δεν συμφωνώ με ε, και να ευχαριστώ μονομανής ε, και επίμονος φανατικός ε, απέναντι σε άλλους σε σχέση με αυτά που είπαν οι προηγουμένοι. Να σας πω ότι γι' αυτό για τις διακοιμάσεις των τιμών ξέρουμε ότι είναι παραδείγμα εχθρός των γεωργών και των νέων γεωργών που διστάζουν να πάνε μακροπρόθεσμα από την εργασία και βλέπουμε πόσο καταραίουν αυτές οι τιμές που λένε οι ειδικοί και ότι δεν υπάρχουν άτομα κάτω από το 35 ετών. Πρόκειται για ένα συναγερμό. Θα πρέπει να να αντιδράσουμε και θα πρέπει να δούμε και μακροπρόθεσμα τι θα γίνει γιατί για μια επένδυση για 20 χρόνια θα πρέπει ταυτόχρονα να καταλάβουμε ότι αυτοί που θέλουν τώρα βραχυπρόθεσμα να επενδύσουν θα πρέπει να έχουν μια σιγουριά μακροπρόθεσμα. Και αυτά είναι λοιπόν και τα δύναμα σημεία αυτά της Επιτροπής που δεν επιμένει ότι θα πρέπει να ρυθμιστούν οι αγορές και πέρα από το φαινόμενο αυτής της κρίσης που υπενθύμησε ο Στέφαν, επίσης είναι οι τρομερές διακοιμάσει των τιμών. Δύσκολα τα πράγματα χρειάζονται μέσα από το δημόσιο να πετύχουμε του απαραίτητους μηχανισμούς. Υπάρχουν και για να το κάνουμε αυτό, να χρησιμοποιήσουμε ότι υπάρχουν και άλλου μέσα δημοσίου. Σε αυτό το πλαίσιο δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο επίση να πετύχουμε μια ιδιαίτερη ισχυρή πλειοψηφία και να δούμε και για τα συμπληρωματικά μέσα που θα πρέπει και θα πρέπει να έχουμε επαναλαμβάνω μια ισχυρή πλειοψηφία για να αντιμετωπίσουμε και το Συμβούλιο. Κατά την άποψη όμω είναι το πρόβλημα υπαριθμών 1 που αντιμετωπίζει σήμερα η Γεωργία, οποιαδήποτε χώρα και αν προερχόμαστε, με οποιαδήποτε παραγωγή, γιατί όποιο είναι ευτυχισμένο σε μια μεριά προκαλεί δυστυχία του αλλού. Βλέπουμε τα δημητριακά προκαλούν μια κρίση και δυσκολίε παντού απέναντι όμω αυτού που παράγουν κρέα και γάλα και καταλαβαίνουμε ότι πάνω σε αυτά τα σημεία θα πρέπει να κεντρώσουμε την προσοχή μας, με διάθεση να μπορέσουμε κάτι να καταφέρουμε, κάτι το συγκεκριμένο, γιατί δεν λέει και πολλά πράγματα αυτό που λέει η Επιτροπή εδώ πέρα και εδώ, εντάξει υπάρχουν 80% θετικά, αλλά το 20% πάντως αυτά αφορούν και δεν ανταποκριθήκαμε σήμερα σε αυτά, δεν δώσαμε μια απάντηση, κάπω να πω ότι λυπάμαι γι' αυτό αυτό ότι είναι μοιραίο που κυμαίνονται τόσο οι τιμέ. Εντάξει, στο Σικάγο καθορίζονται οι τιμέ των Δημητριακών, οι βάρο τη Ευρώπη, αλλά θα πρέπει και εμεί να βαρύνουμε στι αποφάσει τη διεθνή πάνω να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο που φέρνει καταστρεπτικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Μάρκ. Και τώρα ο Τζέιμ Νίκολσον. Uh, thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευθύ εξ αρχή πρέπει να πω ότι είμαστε σε πολύ προώρη φάση μια διαδικασία που θα προσπαθήσουμε να ολοκληρωθεί μέχρι το Μάιο. Στην πορεία θα γίνουν πολλά πράγματα και πολλέ ανταλλαγέ απόψεων. Το πρώτο που θέλω να κάνω είναι να ευχηθώ κάθε καλό στον Άλμπερτ ε, εν ώψη των δυσκολιών που έχει να αντιμετωπίσει. Υπάρχουν τέσσερα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν και τα οποία ε, θα συζητηθούν ε, σε μεγάλη έκταση καθοδόν. Επίσης κάτι άλλο. Εμείς στην Επιτροπή μας πρέπει να δείξουμε τεράστια υπευθυνότητα πέρα της ευθύνης της ε, συναπόφασης που έχουμε. Διότι δεν μπορούμε πλέον ε, να κατηγορούμε την Κομισιόν για αυτά τα οποία πρόκειται να συμβούν. Από εδώ και πέρα θα συνεισφέρουμε και μάλιστα σημαντικά σε αυτά που πρόκειται να συμβούν. Είναι ευπρόσδεκτο επίσης το γεγονός ότι η Κομισιόν ήρθε στην πλευρά των δύο, με το μέρος των δύο πυλώνων, αυτό είναι καλό. Όμως πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μια κοινή γεωργική πολιτική που να λειτουργεί πραγματικά όχι μόνο στη γραφειοκρατία των Βρυξελών αλλά κατά την εφαρμογή της στα κράτη-μέλη και στα πλαίσια των αγροτών που πρέπει να τη χειριστούν. Μια επιλογή που θα επιτρέψει στους αγρότες να, την, έχουν την ευελιξία να εξασφαλίσουν την ποιότητα και τα υψηλά πρότυπα και την ε, επισητιστική ασφάλεια που απαιτείται όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και πέρα από αυτήν. Πρέπει επίσης να λάβουμε το μήνυμα και να το μεταδώσουμε ξεκάθαρα στην κοινή γνώμη. Αυτό συζητούσαμε και σήμερα. Τελικά, τα ωφέλη που θα προέλθουν από μια ισχυρή κοινή γεωργική πολιτική πρέπει να τα, να, τα κάνουμε ε, αντιληπτά. Να μιλήσουμε για την κλιματική αλλαγή, ας πούμε. Εγώ θεωρώ ότι η γεωργία αποτελεί κομμάτι της λύσης των προβλημάτων που θα προκύψουν με την κλιματική αλλαγή, όχι μέρος του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Εδώ πρέπει να συνδυαστούμε και να περάσουμε το μήνυμά μας. Επανειλημμένος δεν το καταφέραμε αυτό. Επανειλημμένος ε, στις αστικές περιοχές πολλοί θεωρούσαν τη γεωργία, ε, τη θεωρούσαν ένα ε, άγωνο πεδίο. Δεν υπάρχει φτηνή τροφή κύριε πρόεδρε. Η καλή τροφή κοστίζει ασχέτως πώς παράγεται. Επίσης είναι κάτι πολύ που με απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την γραφειοκρατία και τις διαδικασίες. Βεβαίως συμφωνώ. Μέχρι, μέχρι σήμερα το μόνο που κάναμε είναι να, να αυξάνουμε τη γραφειοκρατία, τις διαδικασίες, τις δυσκολίες στην εφαρμογή. Η Μαρία ε, η Μέριτ Μαγκίνες είπε ότι όχι θα έχουμε πλέον ε, κόκκινη γραφειοκρατία αλλά θα έχουμε και πράσινη γραφειοκρατία να ακούμε αυτά που μας προτείνονται πράγμα που θα δημιουργεί ακόμα περισσότερα προβλήματα στους ε, παραγωγούς. Επίσης διατρέχοντας την ε, πρόταση. Βλέπω ότι θα γίνει συζήτηση για το τι εστί ενεργός ε, παραγωγός. Αυτό θα διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Και διαρωτώ με αν μπορεί να υπάρξει μία πολιτική βάση της οποία θα αποφασιστεί αυτή η έννοια. Οι, επίσης οι διακυμάνσεις των αγορών αναφέρθηκαν και αυτές. Δεν μπορεί αυτή να εξαφανιστεί τελείω, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει κανείς να κινείται γρήγορα για να εξασφαλίσει ότι δεν θα εξαφανιστεί η παραγωγή. Και αυτό είναι μία από τις δυσκολίες που, που ε, δημιουργεί η διακύμαση των τιμών. Δείτε τι έγινε με το γάλα όταν ε, ε, έγινε η παρέμβαση. Ίσως η Κομισιόν ε, δεν έκανε ολόκληρο θέμα με το γάλα και το βούτυρο το αγόρασε φθηνά και το πούλησε ε, ακριβά. Δεν νομίζω ότι η Ευρώπη έχασε τίποτα, μάλλον κέρδισε από αυτή την όλη περιπέτεια. Επίσης, το μέλλον είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρότατα. Για πάρα πολύ, πάρα πολύ σε πολύ δύσκολες περιοχές, εξαρτώνται από εμά για να εξασφαλίσουμε τα συμφέροντά τους και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η ε, πολλαπλή συμμόρφωση κλπ. είναι ένα κομμάτι της γραφειοκρατίας την οποία ανέφερα και πιστεύω ότι το σύστημα του πώς γίνεται η εφαρμογή έχει σχέση με αυτό. Βρήκα και στη δική μου περιοχή το πρόβλημα τα προβλήματα προκύπτουν σε επίπεδο κράτους μέλους πολύ συχνά, όπου βεβαίως ερμηνεύονται διαφορετικά οι ίδιες διατυπώσεις, τα ίδια έγγραφα των Βρυξελών. Ε, και όλοι κατηγορούν τις βρυξέλλες για τα πάντα. οι εθνικές και περιφερειακές αρχές πάρα πολύ εύκολα ε, στρέφονται κατά των βρυξελών. πρέπει λοιπόν να παρακολουθήσουμε πολύ πιο στενά και προσεκτικά την εφαρμογή αυτών που έχουμε. Και κλείνοντας κύριε Πρόεδρε θέλω να πω το εξής. Θεωρώ ότι η ΚΑΠ, η κοινή γεωργική πολιτική, θα πρέπει κατεξοχήν να είναι πολιτική γεωργική. Δεν μπορεί να είναι περιβαλλοντική πολιτική, ούτε κοινωνική πολιτική. Ίσως πρέπει να έχουμε τέτοια στοιχεία εντός της, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε τίποτα άλλο παρά μια αγροτική βιομηχανία που θα παράγει τις ε, τροφές που απαιτούμε. Ευχαριστώ. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε τον James Νίκολσον. Συνεχίζουμε. Αντιπρόεδρος Νικουλέσκου. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα έπρεπε να σας πω το εξής, ότι ε, θα ήθελα να κάνω σχόλια πάνω σε τρεις πτυχές. Πρώτα απ' όλα, σχετικά με τους γεωργούς τους ενεργούς. Ας μην ξεχνάμε για αυτούς τον στόχο της ΚΑΠ. Ο στόχος είναι παραγωγή τροφίμων. Στη Ρουμανία έχουμε 2,9 εκατομμύρια εκτάρια αχρησιμοποιητής καλλιεργήσιμης γης και σύμφωνα με υπολογισμούς αυτό μας κοστίζει 300 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο. Το ίμιση λοιπόν των πληρωμών των άμεσων που παίρνει η Ρουμανία σήμερα σπαταλάται σε αυτό. Επίσης πρέπει να ορίσουμε τι θα πει νέος παραγωγός, νέος αγρότης για να αποφύγουμε αδικίες. Σαφής ορισμός. Τρίτον, πληρωμές σε μεγάλες εκμεταλλεύσεις και τα όρια που πρέπει να εφαρμόσουμε εκεί. Σωστό, αλλά πρώτα να ορίσουμε τι εννοούμε μεγάλη εκμετάλλευση και πώς μπορούμε να αποφύγουμε μια αυθαίρετη ε, νομική, ε, έναν αυθαίρετο νομικό διαχωρισμό μεταξύ των, του μεγέθων εκμεταλλεύσεων. Τέταρτον, χρειαζόμαστε μία σαφής δομή της γεωργίας αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Άρα λοιπόν ο δεύτερος πυλώνας πρέπει να έχει τα απαραίτητα κονδύλια, τις απαραίτητες πιστώσεις και τη σωστή διαχείριση. Και τέλος, την τελευταία εβδομάδα στο Στρασβούργο συζητήσαμε και είπαμε ότι καμία μεταρρύθμιση ε, δεν θα είναι εφικτή αν δεν απλουστεύσουμε. Διότι αν απλουστεύσουμε ε, απλουστεύσουμε, ε, αν μειώσουμε τις άμεσες πληρωμές πρέπει να, και να απλουστεύσουμε τη διαδικασία. Βεβαίως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Παραγωγών ανέφερε σήμερα την ε, ιδέα περισσότερων πληρωμών, αύξηση των πληρωμών στον πρώτο πυλώνα. Πρέπει να δούμε εάν με τέτοια ιδέα μπορούμε να την υιοθετήσουμε και αν είναι εφικτή μέσα στον πρώτο πυλώνα. Αύξηση στους νέους γεργούς. Πολύ καλά. Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο Νικουλέσκου. Ρέιμερς τώρα. Ευχαριστώ. Θέλω να προσέξετε αυτό που έχω επαναλάβει πολλές φορές. Εάν επιβαρύνουμε τον πρώτο πυλώνα με πολλά καινούργια στοιχεία, θα αυξήσουμε τη γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία σημαίνει χρήματα, κόστος. Και ε, το μόνο που δεν θέλουμε είναι επιπλέον κόστος περισσότερη γραφειοκρατία, περισσότερο κόστος επιβαρύνει τον παραγωγό, λιγότερη ανταγωνιστικότητα στη διεθνή αγορά. Ας μην ξεχνάμε λοιπόν και το, τη σχέση κόστους-οφέλους των εκμεταλλεύσεων. Δεν λέω να μην ε, ε, έχουν ε, κατά νου την ευημερία των ζώων όλους αυτούς τους περιορισμούς και τις προδιαγραφές, αλλά βασικά ενδιαφέρονται να ζήσει η οικογένειά τους. Επίσης, ε, και οι γεωργοί έχουν 24 ώρες στη διάθεσή τους την ημέρα. Εάν πρέπει λοιπόν να διαθέσουν ε, την 25η ώρα της ημέρας για να συμπληρώνουν γραφειοκρατικά στοιχεία, ε, δεν γίνεται. 24 ώρες έχει το το, 24ωρο. Λοιπόν, να μην χάνει και μερικές ώρες ε, ε, γραφειοκρατικά, ειδικά όταν η γραφειοκρατία έχει δημιουργηθεί λόγω πολιτικών συμφερόντων και όχι επειδή χρειάζεται παραγωγικά, διότι έτσι θα χάσει την παραγωγικότητά του. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η γεωργία αποτελεί τον πρωτογενή οικονομικό κλάδο τον οποίο θέλουμε να αναπτύξουμε και όχι να ε, ε, ε, εμποδίσουμε και επιβαρύνουμε. Ήδη δυστυχώς ο πρωτογενής τομέας μειώνεται, συρρυκνώνεται. Έχουμε ένα μεσαίο ε, ε, ε, δευτερογενή κλάδο, ο οποίος επίπεδο μάλλον παραγωγικότητας που αυξάνεται συνέχεια και από πάνω έχουμε τον, το τριτογενή ε, της γραφειοκρατίας. Συμφωνώ με την ανάγκη σαφούς ορισμού νέου παραγωγού νέου γεωργού εδώ μπαίνουμε σε επικίνδυνα νερά, διότι θέλουμε να ορίσουμε ανώτατα όρια, ανώτατες οροφές. Πού θα αρχίσει λοιπόν η εφαρμογή των ανωτάτων αυτών οροφών. Θα βασιστεί στον νέο ορισμό του γεωργού, του νέου γεωργού, του νέου παραγωγού. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι η πραγματικότητα στον αγροτικό τομέα στην Ευρώπη και μάλιστα στις περιφέρειες είναι πάρα πολύ διαφορετική. Διαφέρει <clears throat> και έτσι πώς μπορούμε να με τον πιο δίκαιο σωστό ορισμό για τον νέο γεωργό. Αυτό που ισχύει στην Ιταλία μπορεί να μην ισχύει στη Σουηδία. Επίσης, όταν ζητάμε περιβαλλοντική προστασία ξεχνάμε τις επιπτώσεις. Ε, ένας γεωργός ο οποίος θέλει να εφαρμόσει ένα περιβαλλοντικό μέτρο διότι είναι εφικτό, είναι βιώσιμο μπορεί σε μια άλλη χώρα να μην μπορεί να εφαρμοστεί και να δημιουργεί ζημιά στην διαμόρφωση της αγροτικής πολιτικής πρέπει να έχουμε κατά νου πάντοτε τις διαφορετικές συνθήκες, ε, τις ε, διαφορετικές καταστάσεις που επικρατούν. Διότι σε ένα μέρος φαίνεται κάτι λογικό, σε μια άλλη χώρα όμως είναι παράλογο. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι και σωστή οικονομική διαχείριση και σωστή οικολογική διαχείριση. Ο γεωργός από τη φύση του, από ένστικτο θέλει να προστατεύει τη φύση διότι από τη φύση ζει. Ε, το, να του πούμε λοιπόν να έχουμε πάντοτε μια εχθρική διάθεση έναντι των παραγωγών και να τους λέμε ότι είσαστε πάντοτε αρνητικοί προς το περιβάλλον δεν είναι ούτε σωστό ούτε δίκαιο. Ευχαριστώ. Πολύ καλά. Ευχαριστούμε ε, τον κύριο Ρέμερς Αλμπερτ Ντόρφαντον. Συμφωνώ με όλα αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι πρέπει να σκεφτούμε, να υιοθετήσουμε μία προσέγγιση πέραν των ε, πολιτικών ομάδων και απόψεων. Πολλά λέμε και πολλά είπαμε τις τελευταίες εβδομάδες για μια δίκαιη κατανομή των πιστώσεων στον πρώτο πυλώνα μεταξύ των κρατών μελών. Αλλά θα πρέπει επίσης να δούμε τι συμβαίνει στο εσωτερικό των κρατών μελών. Εγώ προέρχομαι από την Ιταλία. Ε, στην περιφέρεια μου οι άμεσες πληρωμές του πρώτο πυλώνα είναι κάτω από 50 ευρώ ανά εκτάρια. ενώ παραδίπλα ε, οι πληρωμές είναι 400 ευρώ ανά εκτάριο. Δεν μπορούμε να παρακάμψουμε αυτή την πραγματικότητα. Είναι δυσάρεστη, αλλά είναι πραγματικότητα. Και θα πρέπει να τη συζητήσουμε. Στο προτινόμενο μοντέλο της κατανομής του πρώτου πυλώνα, Και στην πρόταση του Επιτρόπου αναφέρεται η ιδέα να διαθέσουμε <clears throat> ένα πρόσθετο ποσό για μειονεκτικές περιοχές. Δηλαδή κάτι το εντελώς καινούργιο. Διότι μέχρι τώρα συζητούσαμε μόνο για την κατανομή ε, των ε, πιστώσεων στο δεύτερο πυλώνα μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης της υπαίθρου. Δεν επρόκειται μια χώρα περισσότερα ή λιγότερα λεφτά. Ό,τι λεφτά είχε για την ανάπτυξη τη υπαίθρου θα έπρεπε να τα διαθέσει. Ωραία. Τώρα, εάν στον πρώτο πυλώνα δεν βρούμε επιπλέον πιστώσει για τι μειονεκτικέ περιοχέ, αλλάζει η κατάσταση και παρουσιάζεται ένα νέο στοιχείο το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει. Μια εντελώ καινούργια διάσταση. Και ε, επ' αυτού δεν λέει τίποτα η ανακοίνωση του, της Επιτροπής. Εν συνεχεία πολλοί συνάδελφοι ανέφεραν τους νέους παραγωγούς. Δεν ξέρω εάν η πρόταση που ακούστηκε χτες να δοθούν περισσότερα λεφτά για τους νέους παραγωγούς μπορεί να εφαρμοστεί, είναι εφαρμόσιμη. Αλλά ούτε αυτό ξε... αποσαφηνίζεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν. Εγώ πιστεύω ότι οι οικονομικές ανάγκες των νέων γεωργών θα αποτελέσουν στο μέλλον ένα πολύ σημαντικό θέμα. Εάν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση όπως τα τελευταία 30 χρόνια, ε, καλύτερα να κλείσουμε το μαγαζί όπως λέμε και να φύγουμε, διότι δεν θα έχουμε πια κανέναν αγρότη. Δεν θα παραμείνει κανένας, είτε νέος είτε μεγάλος. Εάν θέλουμε να προσελκύσουμε ε, και να κινητοποιήσουμε νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τη γεωργία πρέπει να δούμε εάν έχουμε λεφτά και αν τα λεφτά αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε λογικά εύλογα. για τον δεύτερο πυλώνα ακόμα κάτι. Στο πρόβλημα της ε, από γραφειοκρατικοποίησης, δηλαδή της μείωσης της γραφειοκρατίας για μικρές εκμεταλλεύσεις, δεν, δεν πρόκειται απλώς να λάβουν οι μικρές ε, εκμεταλλεύσεις ε, μία επιπλέον βοήθεια. Ε, πρόκειται απλώς για την απλοποίηση της διαδικασίας καταβολής των πληρωμών. Δεν μιλάμε για τίποτα άλλο περίπλοκο, απλούστευση της διαδικασίας άμεσων πληρωμών, ιδίως για τις μικρές εκμεταλλεύσεις, για να μην ε, χάνονται ποσά, σπαταλιώνται λεφτά σε χαρτομάνι, σε, σε, σε σωρούς χαρτιών. Λοιπόν, απλούστευση της ε, γραφειοκρατίας για μικρές μικρές εκμεταλλεύσεις για να μπορέσουν να απαλλαγούν από την αναγκαστική συμπλήρωση εντύπων, γράφων και όλο αυτό το χαρτί το οποίο μαζεύεται. Σε αυτό συμφωνώ. Ευχαριστώ. Πολύ καλά Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να τονίσω ότι ο πρώτος και ο δεύτερος πυλώνας πρέπει σαφώς να είναι διαχωρισμένοι. Αυτό είναι απαραίτητο, διότι διαφορετικά στο μέλλον θα, αρχι... θα, θα δημιουργηθούν κενά στο δεύτερο πυλώνα, ελλείψεις. Και δεδομένου ότι πάρα πολύ ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στον αγροτικό τομέα δεν είναι σωστό εμείς οι ίδιοι να αυτοπυροβοληθούμε, δηλαδή να ζημιώνουμε ήδη τους εαυτούς μας. Γι' αυτό πιστεύω ότι να, να ενισχυθεί οικολογικά, να πρασινίσει περισσότερο ο πρώτος πυλώνας. Ναι, χωρίς όμως επιπλέον γραφειοκρατική επιβάρυνση. Πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την υποστήριξη του αγροτικού προϋπολογισμού στην κοινή γνώμη. Μην ξεχνάμε την έκθεσή μας στην κοινή γνώμη. Ε, θα δεχτούν τον αγροτικό προϋπολογισμό καλύτερα εάν υπάρχουν περισσότερα πράσινα στοιχεία. Ε, χτες ε, που έγινε αυτό το σεμινάριο, αυτή η ακρόαση για τους νέους παραγωγούς συζητήθηκαν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, πόσο ε, αναγκαία είναι η ανάπτυξη της υπαίθρου, πόσο λίγη παραγωγή κάτω των 35 ετών υπάρχουν στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο μη μας τρομάζει. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει να βρούμε σαφείς απαντήσεις σε αυτήν την έκθεση της Κομισιόν ε, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε το θέμα των νέων γεωργών, νέων παραγωγών. Ε, μην ξεχνάμε και τον τομέα της παιδείας κατάρτισης και τη ενίσχυση των επενδύσεων. Στην Αυστρία έχουμε ένα μοντέλο εγκατάστασης, ενός πριν εγκατάστασης. Εάν ένα νέο άνθρωπο αναλάβει μια γεωργική εκμετάλλευση, λαμβάνει ένα πρίμα εγκατάσταση, ε, ε, ένα, ας πούμε, μια κρατική ενίσχυση για να παραμείνει ενεργή η εκμετάλλευσή του και να συνεχίσει να ζει εκεί. Συγκυριέσκη και μετά Η συζήτησή μας για την μεταρρύθμιση της ε, ΚΑΠ έρχεται σε πολύ εύθετο χρόνο. Δεδομένου ότι ταυτόχρονα συζητάμε τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές, ε, τη στρατηγική του 2020, γίνεται η αναθεώρηση του ε, προπολογισμού πολλών πολιτικών και το, ε, την εξέταση υγείας, το health check της ΚΑΠ. Έχουμε μια κρίση στην Ευρώπη, αλλά μας περιμένουν και νέες προκλήσεις. Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι πολύ ιδιαίτερη. Πρέπει λοιπόν να διαρωτηθούμε τι μορφή θα έχει ο προπολογισμός. Αυτό είναι σημαντικό. Το δεύτερο είναι το εξής. Αν θέλουμε αποτελεσματικές λύσεις πρέπει να αναλύσουμε πραγματικά την αγροτική πολιτική το ιστορικό της και τα επιτεύγματά της. Έχει μεγάλα επιτεύγματα, είναι μια πολύ επιτυχημένη πολιτική. Η προηγούμενη επιτυχία της κοινή αγροτικής πολιτικής ε, δείχνει ότι οι προσπάθειές μας πρέπει να συνεχιστούν. Η πολιτική αυτή θα πρέπει να συνεχιστεί. Είναι ένα από τα μεγάλα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Υπήρου μας. Ιδίως δε τώρα σε μια εποχή που έχουμε τόσα πολλά προβλήματα με την προμήθεια ενέργειας κλπ. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια σοβαρή πρόκληση για την ε, επιστημιστική ασφάλεια. Έχουμε μια κληρονομιά, έχουμε την ιστορία. Και τώρα φτάνω στους πυλώνες. Ο πρώτο πυλώνας σημασία έχει, ε, έχει σημασία για τη συγκέντρωση εσόδων και ο δεύτερος πυλώνας αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη με βάση όμως ποιες μεθόδους, ε, με ποιους πόρους και με ποιους κανόνες θα προχωρήσουμε ε, σε κάθε πυλώνα και πώς θα κατανείμουμε αυτούς τους πόρους ε, ανά κράτος μέλος γιατί βεβαίως η κατάσταση διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, από περιφέρεια σε περιφέρεια. Έχουμε μικρούς και μεγάλους κλήρους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι θα πρέπει να στηρίξουμε, τους μικρούς κλήρους, τις μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις. Τι θα γίνει με την ανταγωνιστικότητα οι μεγάλες γεωργικές επιχειρήσεις, οι μεγάλοι κλήροι είναι πλέον ανταγωνιστικοί, ε, είναι μεγαλύτερης εντάσεως παραγωγής και βεβαίως δεν είναι τόσο φιλική προς το περιβάλλον. Πρέπει να βρούμε και μια χρυσή τομή. Ταυτόχρονα πρέπει να διαρρητηθούν οι μηχανισμοί παρέμβασης, ιδίως στον τομέα των σιτηρών, γιατί ε, εκεί, στα Δημητριακά, ε, ο τομέας επηρεάζεται από τη διακύμανση των τιμών. Ένα άλλος, τομέας είναι και τα, ε, ο τομέας των πουλερικών και της αγοράς κρέατος. Όταν θα έχουμε καλές αποδόσεις στα Δημητριακά στο μέλλον θα μπορέσουμε τις ε, καλλιέργειες αυτές να τις χρησιμοποιήσουμε και για την παραγωγή ενέργειας. Και κατακλείδη κύριε Πρόεδρε, η σταθερότητα είναι σημαντική, συμφωνώ, αλλά δεν είναι το παν. Μην ξεχνάμε και τους εξωτερικούς παράγοντες και τις εξωτερικές συνθήκες, το παγκόσμιο χώρο, τις συζητήσεις των ΠΟΕ, τις διαπραγματεύσεις που γίνονται εκεί. Δεν μπορούμε να απομονωθούμε. Αν απομονωθούμε, τότε η ανταγωνιστικότητά μας θα πληγεί. Όλες αυτές οι οδοί, όλες αυτές οι κατευθύνσεις πρέπει να ληφθούν υπόψη ταυτόχρονα. Δεν μπορώ να φανταστώ μια Ευρώπη χωρίς κοινή γεωργική πολιτική. Μια πολιτική που είναι επωφελή στους πάντες ε, και στους καταναλωτές. Η κοινή γεωργική πολιτική είναι ένα είδος πολιτικής υγείας. Καθορίζει την κατάσταση της υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πολιτική αυτή αφορά τους ανθρώπους, ε, ε, έχει σχέση με τους ανθρώπους. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σεχριογιαυσκή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό το έγγραφο είναι μια πολύ καλή βάση συζήτηση για την ΚΑΠ ε, στην επόμενη φάση. Η Λετωνία θεωρεί ότι μία από τις πιο σημαντικές, ε, ε, τα πιο σημαντικά ζητήματα σε αυτό το έγγραφο είναι οι άμεσες πληρωμές το 2013 που θα εξομοιωθούν οι άμεσες πληρωμές μεταξύ των παλαιών και νέων κρατών θα είναι ένα κρίσιμο έτος. Στη Λετωνία οι άμεσες πληρωμές όμως δεν θα εξομοιωθούν, θα είναι ακόμα πάρα πολύ χαμηλές. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη εκτίμηση ανακράτος μέλος. Το είπαμε αυτό ήδη όταν είχαμε την έκθεση του George Lyon και συζητούσαμε την μεταβατική φάση μετά το 2013. Οι Λετονοί παραγωγοί πιστεύουν ότι η μεταβατική αυτή περίοδος που τους δίνεται είναι ανεπαρκέστατη και πάρα πολύ μικρή. Και αν δείτε τα τελευταία χρόνια τι έγινε θα προσέξετε ότι μία ολόκληρη γενιά ε, υπέστη έναν αθέμητο ανταγωνισμό διότι η παραγωγή ε, παραγωγή υφίστανται πιστεύω διακρίσεις λόγω ιστορικού παρελθόντος και υφίστανται τις επιπτώσεις των κρατικοποιήσεων. Δυστυχώς είναι σε δεσμενή θέση λετωνή παραγωγή και θα είναι σε χειρότερη θέση μετά το 2013. Υπάρχει ένας πυλώνας που είναι ε, υπεύθυνο για τις άμεσες πληρωμές και ένας πυλώνας ο οποίος επηρεάζει την ποιότητα της ζωής. Πρέπει να φροντίσουμε και οι δύο να έχουν επαρκή χρηματοδότηση. οι καταβολές, οι άμεσες πληρωμές στους παραγωγούς θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το μέσο όρο στην Ευρώπη το μέσο όρο εισοδημάτων. Πρέπει να εφαρμόσουμε την αναλογικότητα, την αρχή της αναλογικότητας. Αυτή η μεγάλη συζήτηση την οποία κάνουμε για την ΚΑΠ και την μεταρρύθμισή της βλέπουμε ότι επηρεάζεται πάρα υπερβολικά από μια μεγάλη αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές. Αυτό είναι αναμφισβήτητο και στις οικονομίες. Όμως, πρωτεύον θέμα για όλους τους παραγωγούς μας είναι η εξασφάλιση ενός δίκαιου εισοδήματος. Επίσης, ε, μία δίκαιη φορολόγηση όλων των πολιτών μας. Πρέπει και η φορολογία να συμβάλλει σε έναν ε, δίκαιο διεθνή ανταγωνισμό και να μην τους τιμωρεί. Η Λετωνία θέλει να ε, παραμείνουν πολλά στοιχεία της ΚΑΠ ως έχουν. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι πώς θα δημιουργήσουμε και θα συνεχίσουμε να, ε, να βοηθήσουμε να επιβιώσει μία βιώσιμη και αηφόρο αγροτική πολιτική. Λοιπόν, Όλα αυτά που λέμε είναι πάρα πολύ ωραία. Αλλά πρέπει και οι παραγωγοί να έχουν μερικά λεφτά στους λογαριασμούς τους. Δηλαδή ένα ξεπρεπές εισόδημα. Πολλά ακούγονται για την βιοπικιλότητα, το biodiversity. Ε, φτάνει, αρκεί η παρούσα κατάσταση για την εξασφάλιση της βιοπικιλότητας. Ή πρέπει να κάνουμε ορισμένες αλλαγές. ορισμένες αποφάσεις τις οποίες παίρνουμε όχι μόνο βοηθά ε, ε, την επίλυση των κλιματικών προβλημάτων αλλά επιδεινώνει τις κλιματικές αλλαγές. Από τη μία πλευρά θέλουμε περισσότερα προϊόντα που θα ενισχύσουν τη βιοπικιλότητα αλλά ταυτόχρονα βλέπουμε και ζημιές που υφίστανται η παραγωγή. Εάν μπορέσουμε να πείσουμε τους πολίτες της ΕΕ ότι η κοινή αγροτική πολιτική βοηθάει κοινωνικά το δημόσιο συμφέρον, τότε θα μας υποστηρίξουν στις αποφάσεις μας. Δεν συμφωνώ ότι δεν υπάρχει κοινωνική πτυχή εδώ. Δεν, είμαστε απλώς, δεν μοιράζουμε απλώς χρήματα εδώ, αλλά θέλουμε να προβάλλουμε μία θετική εικόνα στη δημοσιότητα ε, και να μας και να πείσουμε τους πολίτες μας ότι προτείνουμε ε, σωστά πράγματα. Από τη σοσιαλδημοκρατική μου άποψη ε, πιστεύουμε ότι το μοντέλο, το μοντέλο μας μοιάζει με ορισμένες προτάσεις που αναφέρει το έγγραφο εδώ μία διαβάθμιση δηλαδή των ε, άμεσων πληρωμών που θα συνδέονται με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια. Το, η δεύτερη βασμίδα πληρωμών ε, προσφέρει περισσότερες πιστώσεις στις μειονεκτικές περιοχές και η τρίτη βαθμίδα προβλέπει επιπλέον ε, πληρωμές για προηγμένες τεχνολογίες που θα εφαρμοστούν οι προηγμένα συστήματα στην γεωργία, στη γεωργική παραγωγή. Ο στόχος του δεύτερου δεύτερου πυλώνα οπωσδήποτε πρέπει να επικεντρώνεται στην ανταγωνιστικότητα και στις καινοτομίες. Με αυτά τα δύο στοιχεία θα ωφεληθούν οι γεωργοί. Δεν μπορούμε εδώ να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση. Πρέπει οι παραγωγοί οι οποίοι ε, καινοτομούν και ε, να αμείβονται και οι ε, ε, φροντίζουν ε, το περιβάλλον, εφαρμόζουν περιβαλλοντικά μέτρα να αμείβονται. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε να δίνονται οι πληρωμές ανάλογα με την γη, με, το στοιχείο της εκμεταλλεύσιμης καλλιεργήσιμης γης. Πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε μία ανεξάρτητη υγιή και βιώσιμη γεωργία να αναπτύξουμε την Ήπεθρο, να μην χάσουμε αποφάσεις, από τα, να μας πάρουν το δικαίωμα αποφάσεων από τα χέρια μας και να φροντίσουμε γενικά την ευημερία των πολιτών μας και των γεωργών. Γι' αυτό ε, τονίζω το κοινωνικό στοιχείο, διότι σε αυτές τις προσπάθειές μας πρέπει να μας υποστηρίξει όλη η κοινωνία. Πολύ καλά. Σας ευχαριστούμε κύριε Ρόντες. Κύριε μετά. Μικρόφωνο παρακαλώ, μικρόφωνο. Μικρόφωνο. Sorry, Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, δύο σημεία. Ο Στίβεν Φολ έφυγε και είχα κάτι να τον ρωτήσω πόσο μικρή πρέπει να είναι η γεωργική επιχείρηση για να θεωρείται ότι δικαιούται την ελάχιστη ενίσχυση. Γιατί διαχωρίζουν, διαχωρίζουν, διαχωρίζουν και τελικά φτάνουμε σε μικρότερο μέγεθος. Τι καλός τρόπος να μπουν νέοι αγρότες. Κάθε φορά που αποκτάνε ένα μωρό, διαιρούν ε, την γη τους και βεβαίως έχουμε ένα νέο αγρότη, επιπλέον ενίσχυση, αλλά κάποιος τα πληρώνει όλα αυτά και δυσανάλογα μάλιστα και δεν θα ε, αργήσουμε να δούμε τους ε, φόρους να ανεβαίνουν. Δεύτερον, ακούσαμε τα περί κλιματικής αλλαγής. Η εκμετάλλευσή μου αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Αγγλία χτες, 30 ε, Νοεμβρίου, καλυπτόταν από, 60, από 6 εκατοστά χιονιού. Αρκετά κάνατε για να σταματήσετε την υπερθέρμανση, αγαπητοί φίλοι. Σταματήστε πια, μην φροντίζετε άλλο. Πολύ καλά. Evans. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένας από τους προλαλήσαντες αναφέρθηκε στις διαφοράς εντός κρατών μελών και όχι ανάμεσα σε κράτη-μέλη εδώ ας πούμε εγώ που εκπροσωπώ την Ουαλία, την εκλογική μου περιφέρεια, αυτό θέλω να το υπογραμμίσω σε σχέση με τις άμεσες πληρωμές που διαφέρουν σε σχέση με τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου. Η παραγωγή και οι ενώσει του στην Ουαλία το βλέπουν τελείω διαφορετικά γιατί αυτέ οι πληρωμέ είναι πολύ σημαντικέ για αυτού. Πάρα πολλοί από αυτού εργάζονται σε ε, λιγότερο ανεπτυγμένε περιοχέ, σε δύσκολε περιοχέ και πολλοί βρίσκονται στα όριο. Πολλοί συνάδελφοι αναφέρθηκαν στι ε, δύσκολε παγκόσμιε ε, συνθήκε στι αγορέ, τι διακοιμάσει των τιμών, την αύξηση των τιμών και το γεγονό ότι του πιέζουν του καλλιεργητέ ε, ε, οι λιανέμποροι και όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στη διατροφική αλυσίδα. Άρα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις άμεσες πληρωμές για να επιβιώσουν οικονομικά. Ξέρω ότι δεν πρόκειται να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση πολύ σύντομα. Έτσι λοιπόν ε, όσον αφορά τη δική μου εκλογική περιφέρεια η κατάργηση των άμεσων πληρωμών θα οδηγήσει σε εξαφάνιση πολλούς παραγωγούς. Θα ήθελα αυτό να το υπογραμμίσω Παραδέχομαι ότι η κοινή γεωργική πολιτική θα περάσει ε, σε άλλου είδους ε, ε, πληρωμές με βάση τις εκτάσεις. Αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται επαρκής μεταβατική περίοδος ώστε να προστατευτούν οι παραγωγοί. Συμφωνώ και με τους άλλους που είπαν ότι χρειάζεται απλούστευση αλλά και περισσότερες λεπτομέρειες για την αλλαγή των πρώτο και δεύτερο πυλώνα για να δούμε και ποιες είναι οι επιπτώσεις τους όμως πρέπει το θέμα της ε, επιστημικής ασφάλειας που βρίσκεται στο επίκεντρο να το συζητήσουμε. Όπως είπαν επίσης πολλοί από τους προλαλήσαντες, υπάρχει και η παραβαλλοντική ευθύνη και ο ρόλος των ε, παραγωγών στην αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θεωρώ ότι τα δύο αυτά θέματα, το θέμα της επιστικής ασφάλειας, της ανάπτυξης υπαίθρου και του περιβάλλοντος και της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής μπορούν να διαχωριστούν από την γενικότερη πολιτική. Ευχαριστώ. Θα ευχαριστήσουμε. Ο κύριος Δανέλης. Grazie, Θα αναφερθώ σε ένα θέμα που θεωρώ ότι είναι κομβικής όμως σημασίας. Νομίζω ότι για την προστασία και την ενίσχυση του ευρωπαϊκού γεωργικού μοντέλου αλλά και την διαχείριση της ευρωπαϊκής υπαίθρου απαιτείται αφενός η στήριξη νέων και δυναμικών στοιχείων στην Ήπεθρο αλλά και η δημιουργία προϋποθέσεων ώστε να μετακινηθούν ή να επιστρέψουν στην Ήπεθρο. Νέοι ε, και δυναμικοί που να μπορούν να ασχοληθούν ε, αποτελεσματικά με την γεωργία. Ε, έτσι η στροφή προς τους ενεργούς αγρότες είναι ορθή. Είναι και μια ευκαιρία να διορθώσουμε μια στρέβλωση τη δημιουργία του φαινομένου του κατεπάγγελμα επιδοτούμενου αγρότη. Ε, πρέπει όμως να αρχίσουμε να συζητάμε για τα κριτήρια με τα οποία θα χαρακτηρίζουμε τους ενεργούς αγρότες, καθώς επίσης και θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά από χώρα σε χώρα, αλλά και από περιφέρεια σε περιφέρεια πιθανώς, μέσα και σε ε, ίδιες χώρες. Παράλληλα νομίζω ότι η συζήτηση για την ε, μεταρρύθμιση της ΚΑΠ είναι μια θαυμάσια ευκαιρία για μας να ανοίξουμε μια συζήτηση και να αποσαφηνίσουμε και μεταξύ μας αλλά και προς όλες τις κατευθύνσεις ότι για τη δημιουργία των προϋποθέσεων της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της διευκόλυνσης της παραμονής στην Ήπεθρο ε, απαιτείται αφενός η μέγιστη συνέργεια μεταξύ των διαρθρωτικών ταμείων στο σύνολό τους αλλά και επίσης για την χάραξη οριζόντιων πολιτικών και κοινοτικών και εθνικών. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία και μια υποχρέωσή μας να ανοίξουμε αυτή τη γενικότερη συζήτηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Λούλινγκ. Ε, ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις 18 Νοεμβρίου, την Πέμπτη, περασμένη, είχα συζητήσει με πολλούς συναδέλφους ότι Σύμφωνο με τις γενικές γραμμές της έκθεσης, αλλά ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Και θα πρέπει να αναλύσουμε κάθε λέξη εδώ πολύ προσεκτικά και να καταστήσουμε σαφές προς ποια είναι η δικιά μας άποψη. Εμπεριστατωμένη λοιπόν ανάλυση του κειμένου χρειάζεται. Έχω πει ότι και με και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να δηλώσουμε σαφώς ότι έχουμε το δικαίωμα μιας κοινή αγροτικής πολιτικής που να καλύπτει όλες τις αγροτικές εκτάσεις σε όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ότι η ζωή και τα εισοδήματα ενός παραγωγού πρέπει να είναι ισοδύναμη και συγκρίσιμα με, τους, με πολίτες που απασχολούνται σε άλλους κλάδους και επιτελούν άλλες εργασίες δεν πρέπει να δεχόμαστε εάν ορισμένοι κλάδοι της οικονομίας ε, υποφέρουν ορισμένα επαγγέλματα ε, να αναλαμβάνουμε εμείς την ευθύνη επειδή συνέχεια κατηγορούν εμάς ότι φταίμε εμείς για όλες τις μιζέριες που υπάρχουν. Οι καταναλωτές βεβαίως επωφελούνται ιδιαίτερα από τις χαμηλές τιμές των προϊόντων Γι' αυτό πρέπει να τους εξηγήσουμε ότι οι άμεσες καταβολές βοηθούν στην επίτευξη ψηλής ποιότητας σε λογικές τιμές, τροφίμων βέβαια και προϊόντων αγροτικών. Τώρα, αν έχω καταλάβει καλά τον Επίτροπο, θέλει να πρασινίσει περισσότερο η ΚΑΠ γιατί λέει ότι εάν πρασινίσουμε περισσότερο την ΚΑΠ μπορούμε να πουλήσουμε καλύτερα τις πιστώσεις προς την ΚΑΠ και ότι μπορούμε να πουλήσουμε καλύτερα στη δημόσια γνώμη τις δαπάνες. ωραία αυτή η ιδέα, δεν λέω, αλλά να είμαστε σαφείς. Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτής της πρότασης και συμφωνώ απόλυτα με τους προλαλήσαντες συναδέλφους. Πρέπει να είναι σαφέστατο ότι αυτή η πιο πράσινη ΚΑΠ, τα επιπλέον πράσινα στοιχεία, θα έχουν σαφή επίπτωση στα εισοδήματα των παραγωγών. και δεν, μπορούμε, δεν, δεν πρέπει να οδηγήσουν στο να ανθεί περισσότερο ακόμα η γραφειοκρατία χτες όταν ε, συμμετείχα στη συζήτηση που έγινε χτες με τους, για τους νέους αγρότες μίλησα και με την αντιπροσωπεία του Λουξεμβούργου και μου είπαν ότι δεν είναι δυνατόν να επιβαρύνουμε με περισσότερη γραφειοκρατία τους παραγωγούς από ότι ήδη επιβαρύνθηκαν με την πολλαπλή συμμόρφωση, το cross compliance. Και δεν μπορεί τώρα αυτή η τα πράσινα στοιχεία να μπουν όλα στον πρώτο πυλώνα γιατί περισσότερα λεφτά δεν θα πάρουμε. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνουν τα στοιχεία αυτά στο δεύτερο πυλώνα και εάν υπάρξει θέμα αποζημιώσεων των παραγωγών θα πρέπει οι αποζημιώσεις των μειονεκτικών περιοχών όπως είπε ο κύριος Ντόφμαν ήδη να παραμείνουν συγγνώμη στη δεύτερο πυλώνα. Στο δεύτερο πυλώνα. Uh, είχα συμμετάσχει σε αυτό το φόρουμ με τους νέους παραγωγούς και αναρωτιέμαι αυτή η κυρία Εμπειρογνώμων η οποία μας παρουσίασε την ομιλία της εχθές πόσο πληρώθηκε εγώ δεν κατάλαβα γρήγορα από αυτά που μας είπε η κυρία αλλά Καλό είναι πρόεδρε να προσέχουμε στους εμπειρογνώμονες αναθέτουμε τέτοιες παρουσιάσεις γιατί τέτοια τρελά πράγματα που άκουσα χτες από την ε, λεγόμενη ειδική, εμπειρογνώμονα, δεν έχω ξανακούσει ποτέ. Ε, βγάλαμε, εμείς πετάξαμε τα ακουστικά μας και τα μικρόφωνα. Λοιπόν, προσέξτε παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, τα πολύτιμα κονδύλια της Επιτροπής μας να δαπανώνται καλύτερα και σε ε, καλύτερες εμπειρογνώμονες από αυτήν που ακούσαμε χτες. Όσον αφορά τώρα την εισαγωγή των ορίων για τις άμεσες πληρωμές σε, σε παραγωγούς, δραστήριους παραγωγούς δηλαδή, προσέξτε, προσέξτε τις καταχρήσεις. Είναι πάρα πολύ εύκολο να παραβιάσει κανείς ένα τέτοιο ανώτερο όριο, μια οροφή διότι μπορεί να μοιράσει κανείς μία εκμετάλλευση στα παιδιά του, στη γυναίκα του, σε διάφορα τεμάχια για να έχει απαιτήσει ε, για τις πληρωμές αυτές και να παρακάμψει την οροφή. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε μία ισχυρή πλειοψηφία σε αυτή την Επιτροπή για να περάσουμε τους στόχους μας. Και για να επιβιώσει και αναπτυχθεί μια δίκαιη αγροτική πολιτική. Ευχαριστούμε την κυρία Λούλινγκ. Να σας διαβεβαιώσω για την εργασία των εμπειρογνωμόνων ότι εκεί όλοι μαζί λάβαμε αυτή την απόφαση. Δεν ήταν αποκλειστικά δική μου. Ashworth. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ε, ε, αυτή η επιθυμία για μια ισχυρή στήριξη της κοινής αγροτικής πολιτικής ε, ε, ε, οφείλεται σε ένα στατιστικό στοιχείο που δεν έχω ξεχάσει ότι αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι της χώρας μου δαπανούν 11% του διαθέσιμου εισοδήματός τους σε τρόφιμα. Το μέσο εισόδημα του μέσου ε, παραγωγού είναι το 50% του, μέσου, ε, του εισοδήματος του μέσου Ευρωπαίου. Δεν μπορεί να τα έχουμε όλα λοιπόν. Ε, δηλαδή το αντίθετο ύπαρξη μιας κοινή αγροτικής πολιτικής θα διεπλασίαζε τις δαπάνες για τρόφιμα και αυτό θα είχε κακό αποτέλεσμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω όμως να είμαι επιφυλακτική. Και η επιφύλαξή μου έχει σχέση με τον προπολογισμό. Δηλαδή, για να σας το δείξω, μέχρι στιγμής αυτό που βλέπουμε ε, από την Κομισιόν όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις είναι ένας κατάλογος επιθυμιών. Ε, ε, αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο προϋπολογισμός, χρειαζόμαστε περισσότερη σαφήνεια όσον αφορά τους αντικειμενικούς σκοπούς. Αντιλαμβανόμαστε την επιθυμία της, της Κομισιόν για θέματα να γίνει πιο πράσινη η κοινή αγροτική πολιτική, να φύγουμε από την ιστορική κοινή αγροτική πολιτική και να έχουμε την έννοια του ενεργού ε, παραγωγού. Αλλά όλα αυτά μου φαίνονται περαιτέρω επιπλοκές, περισσότερη γραφειοκρατία και προσθήκη επιπλέον κόστους στον κλάδο που για μένα σημαίνει ότι κινούμαστε σαφώς προς την ε, λάθος κατεύθυνση. Αυτό που είναι σαφές είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση για την ε, κοινή γεωργική πολιτική ακόμα και με τις υφιστάμενες δομές γιατί η, ανάγκη για καλύτερη κατανομή θα σημαίνει ότι θα υπάρχει ανάγκη για περισσότερη, περισσότερη ίση μεταχείριση των κρατών μελών και αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν μεγαλύτερες απαιτήσει από τον προπολογισμό. Όμως προειδοποιώ, ο, αυτός ο προπολογισμό έτσι κι αλλιώς θα είναι ε, μικρότερος και από δημοσιονομική σκοπιά αυτό το οποίο παν, παντού χρειαζόμαστε κυρίως κυρίω όμω στο πλαίσιο τη ε, κοινή γεωργική πολιτική είναι μεγαλύτερη ευελιξία, δυνατότητα να αντιδράσουμε και να ανταποκριθούμε στι περιστάσει καλύτερα. Και αυτό υπήρξε πάντα αδυναμία του συστήματο, ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Κυρίω με μικρότερο προπολογισμό, η δυνατότητα ευελιξία εντό του προπολογισμού αυτού είναι πάρα πολύ σημαντική. Τα επισημαίνω αυτά, διότι ω και ε, μέλο τη Επιτροπή ΣΟΡ, η οποία εντοπίζει την ε, μεταρρύθμιση του συνολικού προπολογισμού, πρέπει να πω ότι εκεί οι εισηγητές έχουν ε, προτείνει τρεις προτάσεις για την αναδιοργάνωση των έξι τίτλων του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού. Δύο από αυτές τις προτάσεις ε, προβλέπουν ε, η κοινή αγροτική πολιτική να ενταχθεί μαζί με τα θέματα ενέργειας και κλιματικής αλλαγής. Άρα, εγώ ανησυχώ ότι αυτή τη στιγμή η κοινή αγροτική πολιτική είναι το 42% του προπολογισμού. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι βεβαίως θα αντιμετωπίσει πρόβλημα εδώ θα υπάρχει θέμα και γι' αυτό κάνω μια έκκληση μεγαλύτερη, ε, ε, να επικεντρωθούμε καλύτερα στο σκοπό που επιδιώκουμε. Δεν είναι ούτε κοινωνική, ούτε χωροταξική, ούτε περιβαλλοντική πολιτική. Είναι ε, αγροτική πολιτική. Δεν υπάρχει αρκετή έμφαση και αυτό την αποδυναμώνει. Η ουσία, το θετικό σημείο της κοινή γεωργικής πολιτικής είναι ότι είναι μια πολιτική τροφίμων, ότι υπάρχουν 500 εκατομμύρια άνθρωποι που μπορούν να υποφεληθούν από αυτή. Όχι μόνο 5 εκατομμύρια μέσα στο λόγο του ότι είναι μια γεωργική πολιτική. Άρα εγώ ζητώ μεγαλύτερη έμφαση στο σκοπό μας και καλύτερη στόχευση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ευχαριστούμε κύριε Άσουορτ. Όλοι μας θα πρέπει να καταβλάμε αυτή την προσπάθεια να εξηγήσουμε ότι δεν είναι μόνο πολιτική για τους Ευρωπαίους γεωργούς, αλλά για όλους τους πολίτες η ΚΑΠ. Έτσι μόνο θα μπορέσουμε να έχουμε και την υποστήριξη όλων ε, και στο Κοινοβούλιο. Πατράνε Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, να σας πω ότι η ανακοίνωση της Επιτροπής κατά γενικό τρόπο εντάξει συμφωνώ Ταυτόχρονα όμως με ανησυχεί, με ανησυχεί πολύ. Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα γι' αυτό να χρησιμοποιήσω μια έκφραση. Έχουμε ένα όμορφο κουτί. Όμορφο. Και εκεί να βάλουμε το χριστουγεννιάτικο δώρο. Και αυτό ωραίο δωράκι. Α, τι γίνεται, εδώ πέρα έχουμε μόνο το άδειο κουτί. Δεν ξέρουμε τι θα βάλουμε μέσα σαν δωράκι μέσα σε αυτό το ωραίο κουτί. Θα το σκεφτούμε αργότερα ποιο θα είναι το δώρο. Λοιπόν, εγώ ανησυχώ ιδιαίτερα το τι θα βάλουμε μέσα σαν δωράκι, τι θα διαλέξουμε. Εντάξει, η παρουσίαση είναι όμορφη απ' έξω, η συσκευασία υπέροχη. Ορισμένοι ήθελαν ε, να αλλάξουν την αρχιτεκτονική της ΚΑΠ και είχε προταθεί στην Επιτροπή να φύγουν από τη μέση οι πυλώνες, ε, να έχουν είτε να έχουμε τρεις αντί για δύο πυλώνες. Τέλος πάντων, ε, χαίρομαι που η Επιτροπή δεν αφέθηκε να πιστεί και διατήρησε τους δύο πυλώνες. Και εντάξει, όταν μιλάμε για τα δημόσια ε, αγαθά λέμε ότι υπάρχουν πρώτης γενιάς, δεύτερης γενιάς και υπερίσχυσε αυτή η άποψη και στην ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρεται ότι ο κύριος στόχος της ΚΑΠ είναι να βγάλεις την παραγωγή προϊόντα, τρόφιμα ποιοτικά και να είμαστε σίγουροι. Υπάρχει μια εγκύμηση γι' αυτό. Εδώ το ξέραμε όλοι λοιπόν, αλλά από την άλλη μεριά όμως υπήρχαν δυνάμεις που θα ήθελαν να αλλάξουν τα πράγματα και χαίρομαι εγώ που τα πράγματα παρέμειναν ως έχουν. Υπήρχαν διάφοροι που ήθελα να ξεχάσουμε το ουσιαστικό, το κύριο σημείο της γεωργίας και αναφέρομαι κυρίως σε περιβαλλοντικά κινήματα που άσκησαν ιδιαίτερη πίεση και η ΚΑΠ όλα ένα και γινόταν κάτι που είχε να κάνει με την οικολογία. Θα πρέπει να μην ξεχνάμε όλα αυτά στα οποία έχουμε πρόσβαση και να δούμε και την τελική έκδοση της Επιτροπής. Καταλαβαίνουμε ότι ε, όλο και περισσότερο ρόλο παίζει η συνιστόσα περιβάλλον. Κάτι που δεν θα πρέπει όμως να ξεχνάμε. Μιλάμε για την κοινή γεωργική πολιτική και όχι για μια περιβαλλοντική κρυμμένη πολιτική. Έχει θέση της ε, αλλού η περιβαλλοντική πολιτική. Εδώ μιλάμε για γεωργική πολιτική. Και όταν μιλάμε για τη συνιστόσα αυτή την οικολογική, να απευθύνω ερώτημα στην Επιτροπή. Μιλάμε για την κλιματική αλλαγή. Μιλάμε τόσο για το θέμα αυτό. Ένα θέμα όμως που στη συνέχεια δεν αναπτύσσεται περισσότερο και έτσι κάποιος ε, σχηματίζει την εντύπωση ότι τελικά η γεωργία θα παίξει, θα παίξει τον πρώτο ρόλο κατά της κλιματικής αλλαγής. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια πρόθυσε διάφορες ενέργειες περισσότερο από άλλους τομείς και αυτό για να δώσει τη μάχη της κατά της κλιματικής αλλαγής. Αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο ο γεωργικός τομέας να αναλάβει το έργο αυτό. Και ακόμη σχετικά με την συνιστόσα την οικολογική. Κάτι που με ανησυχεί πώς θα πετύχουμε μια ισορροπία ανάμεσα σε μια πιο πράσινη γεωργία και στον προϋπολογισμό που βλέπουμε ότι δεν παίρνει περισσότερα κονδύλια. Ταυτόχρονα και με την ανάγκη ότι θα πρέπει να απλουστεύσουμε τα πράγματα. Όλα αυτά έχουν σχέση μεταξύ τους. Για να δούμε πώς το δίλημα αυτό θα το λύσουμε. Αυτό με, αυτά με απασχολούν. Δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω περισσότερα, αλλά να σας πω κάτι που για μένα από την Πορτογαλία και από μια ε, ιδιαίτερα απομακρυσμένη περιοχή της Αζόρας, αυτά τα θέματα έχουν ιδιαίτερη σημασία. Μιλάμε για την προστασία των μικρών καλλιεργητών αλλά ποιοι είναι οι μικροκαλλιεργητές και οι μικροκαλλιέργειες, ποια είναι τα κριτήρια για αυτούς, γιατί εκεί δεν συμφωνούμε όλοι. Πώς θα έχουμε τον ορισμό του μικροκαλλιεργητή και μιλάμε επίσης για μειονεκτικές περιοχές και την υποστήριξη σε αυτές. Αλλά οι περισσότερες ενισχύσεις είναι στα πλαίσια του δεύτερου πυλώνα που σημαίνει συγχρηματοδότηση. Και όταν μιλάμε για συγχρηματοδότηση από τη στιγμή που δίνουν τη μάχη του τα κράτη-μέλη κατά τη, βα... της βαθιάς κρίσης του προπολογισμού, τι σημαίνει ότι οι μενεκτικές περιοχές ε, θα έχουν ε, πάντα τα χάλια τους, ε, δηλαδή θα παραμείνει η κατάσταση ως έχει. Αυτά λοιπόν. Θα ήθελα να ολοκληρώσω και να προσθέσω ότι για μένα το σημαντικό είναι το δωράκι που θα πρέπει να βάλουμε στο κουτάκι μας θα είναι μια κάποιο δίκαιη. Τι σημαίνει όμως να μια μεριά πιο δίκαιη κοινή γεωργική πολιτική. Μια κατανομή, ένα εκτάριο που θα μεταβάλει σε δικαιότερη πολιτική την ΚΑΠ και μετά τους ε, δίκτες προσαρμογής. Τι θα είναι, θα είναι παιδικά παιχνιδάκια, θα ε, βάλουμε κάτω τις καρτούλες μας και η κατανομή θα είναι όπως πριν. Όλοι κάνουν τους λογαριασμούς τους. Αλλά αν τελικά με τους λογαριασμούς αυτός ο διορθωτικός συντελεστής ε, παίξει αυτό το ρόλο. Αυτοί που παίρνουν τα περισσότερα παίρνουν πάντα περισσότερα και αυτοί που παίρνουν λιγότερα θα παίρνουν τα λιγότερα, τότε τίποτα δεν θα μεταβληθεί. Ελπίζουμε η Βασίλισσα ενός άλλου είδους δώρο να μας φέρει. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ο Βασίλης μας έφερε σαν δωράκι την ε, συνήθεια της Αβώνας. Άρα λοιπόν έχουμε την ευθύνη να τα προχωρήσουμε όλα αυτά. Εμείς είμαστε εκείνοι που θα τα κάνουμε. Γκίνες. Ε, λοιπόν και ολοκληρώνουμε έτσι. Thank you. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ελπίζω να μην ε, μου αναθέτεις όλη την ευθύνη επειδή είμαι η τελευταία ομιλήτρια. Όμως ε, αυτά που είπαμε σήμερα το πρωί μεταφέρονται και σήμερα το απόγευμα. Συμφωνώ ιδιαίτερα με αυτά που είπε ο Ρίτσο Ντάσουαρτ σε σχέση με το αγροτικό εισόδημα και την σημασία τη παραγωγή τροφίμων. Δεν άργελε στου καταναλωτέ τη Ευρώπη το γεγονό ότι υπήρχε έλλειψη τροφίμων και ανέβηκαν οι τιμέ. Δεν θα πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη που έχουμε αυτή την πολιτική που προσφέρει ποιοτικέ τροφέ στου καταναλωτέ μα. Η Κομισιόν προσπαθεί, ε, πρέπει να δικαιολογήσει. Δεν είμαστε σε θέση ισχύω αυτή τη στιγμή, είμαστε σε αμυντική θέση. Ε, επίσης προέρχομαι από τον προπολογισμό και ασχολούμαι με τον προπολογισμό του επομένου έτους. Υπάρχουν και εκεί ανησυχίες. Τελικά προσπαθούμε να ταιριάξουν οι ιδέες μας μέσα σε, στα κάποια ποσά. Αυτό είναι ακριβώς αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε. Φοβάμαι όμως ότι ακριβώς αυτή η συζήτηση γίνεται σήμερα το απόγευμα. Θα θέσω κάποια ε, ερωτήματα. Ο Επίτροπος έχει τρία ερωτήματα στο έγγραφο, αλλά ένα έχει επιλεγεί. Αν είμαστε πραγματικά ειλικρινείς ε, ως πολιτικοί, χρειαζόμαστε ε, πληροφορίες και για τα τρία. Χρειαζόμαστε τις επιπτώσεις, ποιες είναι οι, θα είναι οι επιλογές μας και πώς θα επηρεάσουν τους παραγωγούς και την παραγωγή τροφίμων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι πληροφορίες δεν μας δίνονται. Τώρα, όσον αφορά την ισότητα, την δικαιοσύνη, Πολύ σωστό ερώτημα. Ο, καθένας που έχει παιδιά θα ξέρει ότι κανένας δεν θεωρεί ότι αντιμετωπίζεται με δικαιοσύνη. Κάθε παιδί σου προσπαθεί ε, να, να αποδείξει ότι ε, εσύ ευνοείς τα άλλα, ότι είσαι άδικος απέναντί του. Έτσι δεν είναι. Ε, είναι πολύ δύσκολη αυτή η αντίληψη και νομοθετικά. Επίσης τώρα οι πληρωμές με βάση τις ε, εκτάσεις. Ε, αν βάλω το καπέλο ειδικού, αυτές πιστεύω ότι θα αυξήσουν το κόστος παραγωγής, είναι εμφανής, γιατί αφορούν τις τιμές ας πούμε ε, νοικίασης της γης. Ας δούμε ποιες θα είναι αυτές οι επιπτώσεις αυτού του συστήματος. Με κάποιο μέγιστο ποσό, ναι, θα αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες κάποιων που φοβούνται για πολύ μεγάλες ε, πληρωμές σε κάποιους παραγωγούς. Αλλά ίσως κάποιοι παραγωγή ε, αξίζουν αυτές τις πληρωμές αν έχουν μεγάλη ε, δραστηριότητα. Ε, άρα είναι δύσκολα αυτά τα θέματα για να τα νομοθετήσουμε και χρειάζονται μια περισσότερο σε βάθος συζήτηση από αυτήν εδώ για το πώς θα επηρεαστεί η παραγωγή τροφίμων που είναι και η ουσία αυτής της συζήτησης. Το θέμα των ενεργών παραγωγών. Θεωρώ ότι αυτοί πρέπει να είναι αυτοί που θα υποφεληθούν. Σε κάποια κράτη-μέλη είναι πιο σαφές ότι αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι πληρώνονται. Πρέπει να δούμε πού υπάρχουν τα προβλήματα στα κράτη-μέλη, είναι, ποιες είναι οι περιπτώσεις που τα χρήματα δεν πηγαίνουν στους ε, ενεργούς αγρότε και πηγαίνουν στα γήπεδα γκολφ και αλλού. Γιατί πρέπει ακριβώς να εντοπίσουμε το πρόβλημα και να δούμε ποιο είναι αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει και το ευρύτερο θέμα που έχω θέσει στη δημόσια διαβούλευση. Τι σημαίνει ε, δραστήριος ενεργός παραγωγός είναι αυτός που ασχολείται με πλήρη απασχόληση, είναι κάποιος που διδάσκει αλλά ασχολείται και με την παραγωγή. Είναι δύσκολα ζητήματα τα οποία ενδεχομένως να αποφεύγουμε. Αλλά δεν πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να μιλήσουμε ξεκάθαρα για όλα αυτά για να λάβουμε σωστές αποφάσεις επίσης θεωρώ ότι αυτό το οποίο είπα για το πρασίνισμα του, πράσινου πυλώνα, του πρώτου πυλώνα εξακολουθούν να ισχύουν. Ανησυχώ για την ε, υπερβολική ρύθμιση του κλάδου ε, ανησυχώ για την υπερβολική έμφαση στις άμεσες πληρωμές χωρίς να υπάρχει επαρκής έμφαση στις αγορές. Αν δεν δούμε την αγορά και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να στείλουμε καλύτερες τιμές ή καλύτερες αποδόσεις στους παραγωγούς θα βλέπουμε μόνο το ένα σκέλος της υπόθεσης. Μην, μην αγνοήσουμε λοιπόν τη στήριξη αγοράς, τη ρύθμιση της αγοράς γιατί όλα αυτά έχουν σχέση με τα θέματα της επιστημιστικής ασφάλειας που μας ανησυχούν βαθιά. Επίσης ε, έγινε αυτός ο γύρος συζητήσεων. Δεν είμαι βεβαία ότι έχουμε ε, χωρίσει περισσότερο σε βάθος από ό,τι την πρώτη φορά και μόνο όταν θα έχουμε την νομοθετική πρόταση της Κομισιόν θα μπορέσουμε να μπούμε στην ουσία αυτής της συζήτησης. Ιδάλλως φοβάμαι ότι η έκθεση θα προσπαθήσει να αποσπάσει κάποιες από τις λεπτομέρειες. Δεν θα με ικανοποιεί όμως η κατεύθυνση των μεταρρυθμίσεων ακριβώς για τους λόγους που σας εξέθεσα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους πήραν το λόγο. Αγαπητέ Διευθυντή Τάσο, 18 παρεμβάσεις είχαμε, απόψεις, διαφορετικές ευαισθησίες, αλλά όλοι συγκλίνουν προς μια ισχυρή ρωμαλαία ΠΑΚ που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και των γεωργών και των πολιτών. Να δώσουμε το λόγο τώρα στον Τάσο Ανιώτη από την Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Γεωργίας. Έχεις το λόγο Τάσο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους για τις πολύτιμες παρατηρήσεις σας αλλά και για τη δουλειά που κάνατε με τον κατάλογο των ερωτήσεων. Δεν νομίζω ότι αυτές οι 74 ερωτήσεις εξαντλούν όλα τα πιθανά ερωτήματα που θα μπορούν να τεθούν και ελπίζω με αυτά που θα πω να μην προκαλέσω περισσότερες ερωτήσεις. Εν πάση περιπτώσει, θα προσπαθήσω να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις και να διευκρινίσω κάποια στοιχεία της ανακοίνωσης, όχι σε σχέση με τις συγκεκριμένες προτάσεις που πρόκειται να γίνουν. Αυτές θα γίνουν αργότερα, όπως γνωρίζετε, αλλά σε σχέση με το πού βρισκόμαστε τώρα σε σχέση με αυτή την ανακοίνωση. Ξεκινάω με αυτό που ακούστηκε ότι πρόκειται για έναν κατάλογο επιθυμιών. Πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι για το τι εστί αυτή η ανακοίνωση, περί τίνος πρόκειται. Ανταποκρίνεται στη δημόσια συζήτηση που έχει γίνει με πρωτοβουλία του Επιτρόπου μας για να δούμε ποια είναι η άποψη της ευρύτερης κοινής γνώμης για την κοινή γεωργική πολιτική. Σαφώς δεν έχουμε απαντήσει ε, για όλα σε όλα τα ερωτήματα. Ξέρουμε όμως πολύ περισσότερα για τις κατευθύνσεις και για τους τομείς όπου υπάρχουν απαντήσεις, ενώ άλλους, για τους τομείς που πρέπει να βρεθούν απαντήσεις. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για που υπάρχουν, υπάρχει σύγχυση και όπου υπάρχουν τρεις εναλλακτικέ. Μία σαφώς την προτιμούμε, αλλά και οι τρεις είναι πραγματικές, οι οποίες διεφάνισαν και από την δημόσια συζήτηση. Η πρώτη εναλλακτική μελετά τις πιθανές επιπτώσεις της ανακατανομής της ενίσχυσης και ε, ε, λαμβάνει υπόψη αυτές τις σημαντικές επιπτώσεις σε κάποιους τομείς και κάποιες περιφέρειες και θεωρεί ότι αυτές οι επιπτώσεις είναι αρκετά ε, σημαντικές και ενδεχομένως εκεί θα πρέπει να σταματήσουμε. Δεν ξέρω αν θα την επιλέξουμε αυτήν ή όχι, πάντω είναι αυτή που ε, συζητήθηκε ευρύτατα. Το ίδιο ισχύει και για την τρίτη ε, εναλλακτική. Δικατοπτρίζει ε, ιδέε που προέρχονται μόνο από μερικά κρατημέλη αλλά και κάποια think tank που έχουν κάνει σοβαρές αναλύσεις. Θα γίνει μια λεπτομερέστατη μελέτη επιπτώσεων και των τριών εναλλακτικών με μια με δύο άλλε εναλλακτικέ. Τι θα γίνει αν δεν αλλάξει απολύτω τίποτα και τι θα γίνει αν τα καταργήσουμε όλα. Γι' αυτό έχουμε ήδη ε, αποτελέσματα. Τώρα, η διαδικασία για τη μελλοντική μεταρρύθμιση της ΚΑΠ έχει ήδη ξεκινήσει. Μία διατμηματική περιοχή ε, με 50 άτομα που συνεδριάζουν. Έχουμε κάνει 7 ε, συνεδριάσεις. Αναλύουμε τις εναλλακτικές. Στις 23 Νοεμβρίου στείλαμε ένα έγγραφο διαβούλευση με τη μελέτη επιπτώσεων, με πιο συγκεκριμένα ερωτήματα και καθορισμό προβλημάτων για το που θέλουμε να πάμε και ζητήσαμε από ε, το την κοινή γνώμη να μας στείλει ε, μέχρι τις 25 Ιανουαρίου απαντήσεις. Τώρα, όσον αφορά τα ερωτήματα που θέσατε, τα περισσότερα από αυτά αφορούν την σχέση πρώτου με δεύτερο πυλώνα και τις άμεσες ε, απευθείας πληρωμές. Πρέπει όμως να ξεκινήσουμε, να καθορίσουμε κάτι ξεκινώντας από τον τίτλο της ανακοίνωσης. Μιλά για τρόφιμα, για το περιβάλλον και για τις εκτάσεις. Και τα τρία αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής. Πουθενά δεν δημιουργούμε την εντύπωση ότι η η κοινή γεωργική πολιτική δεν αφορά την παραγωγή. Αλλά δεν, είναι μόνο, δεν αφορά μόνο την παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Από καιρό τώρα λέμε ότι η γεωργία δεν αφορά μόνο την παραγωγή τροφίμων, αλλά την παροχή υπηρεσιών, κυρίω αγροπεριβαλλοντικών υπηρεσιών που γίνονται όλο και πιο σημαντικέ στο υφιστάμενο πλαίσιο των μεγάλων προκλήσεων. Προσπαθούμε να διευκρινίσουμε τη σχέση πρώτου με δεύτερο πυλώνα, επειδή δεν θέλουμε τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα του δεύτερου πυλώνα να μεταφερθούν στον πρώτο πυλώνα. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Πάντοτε θα υπάρξει ανάγκη να υπάρχουν στοχευμένα μέτρα που ε, προσπαθούν να βελτιώσουν την, ε, το περιβάλλον στο, μέσω της γεωργίας. Είναι συγκεκριμένα, μερικά από αυτά συγκεκριμένα σε τοπικό επίπεδο και μόνο τα κράτη-μέλη μπορούν να καθορίσουν τις προτεραιότητες και να επιδώσουν αυτά τα μέτρα να τα κάνουν να λειτουργήσουν. Εδώ τι επιδιώκουμε. Κάποια απλά μέτρα που ήδη υφίστανται, πολλά από αυτά είναι κομμάτι της καλής γεωργικής περιβαλλοντικής κατάστασης κάποιων κρατών μελών και θέλουμε να ε, βελτιώσουμε το καλό δημόσιο αγαθό που προέρχεται είτε πρόκειται για περιβαλλοντικά ε, περιβαλλοντικό ε, περιβαλλοντική αγρανάπαυση είτε για μια σειρά από άλλα μέτρα είναι μέτρα γνωστά στους παραγωγούς από τη μια πλευρά μας λέει ότι μπερδεύουμε περισσότερο τα πράγματα και από την άλλη πλευρά μας λένε ότι τώρα προτείνουμε να, να ε, αποζημιώσουμε τους παραγωγούς για αυτό το οποίο ήδη κάνουν. Η πραγματικότητα η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε το ειδικό τύπο μέτρων, συνθήκων και περιοχών που πρέπει να εφαρμοστούν αυτά, έχοντας πάντοτε κατά νου ότι δεν θα πρέπει να να περιπλέξουμε έτσι περαιτέρω τα πράγματα, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο γενικότερος στόχος των άμεσων πληρωμών δεν είναι μόνο η παροχή εισοδηματικής στήριξης, αλλά η παραγωγή κάποιων υπηρεσιών και δημοσίων αγαθών που είναι απαραίτητα. Υπάρχουν ήδη κάποιες περιοχές με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Το έχουμε λάβει υπόψη. Φυσικές, φυσικοί περιορισμοί, ότι όπως θέλετε πείτε το. Δίνουμε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να το λάβουν αυτό υπόψη όταν ανακατανέμουν ε, τη στήριξη εντός κρατών μελών. Τώρα, όσον αφορά τα θέματα που αφορούν τους μικρούς παραγωγούς, τους ενεργούς παραγωγούς, τα τα ανώτατα κλπ. Είναι θέματα που αντιμετωπίζουμε και εμεί. Τα θέσατε εσεί τα αντιμετωπίζουμε και εμεί. Το θέμα του ενεργού παραγωγού έχει πάρει μια εντελώς διαφορετική διάσταση από την ώρα που έγινε αποδέσμευση. Γιατί προσφέρουμε όχι μόνο για τα τρόφιμα αλλά και για τις γεωργικές υπηρεσίες και πρέπει, που υπάρχει διαχωριστική γραμμή, πρέπει να απαντηθούν όλα αυτά τα ερωτήματα και μερικές από τις απαντήσεις αυτές δεν έχει άμεση σχέση με το πώς θα καθοριστεί η έννοια του μικρού παραγωγού. Ίσως αυτός να μην είναι ο πάρα πολύ μικρός παραγωγός, ένας ενεργός παραγωγός. Ίσως η λύση σε αυτό είναι πολύ εύκολη, αλλά άλλα ζητήματα είναι πιο δύσκολο να λυθούν. Υπάρχει κοινό, ας πούμε, ε, ορισμός μεταξύ του μικρού παραγωγού ή του ενεργού παραγωγού στα κράτη-μέλη. Ε, τι, τι συνδυασμό ε, ζητημάτων θα κάνουμε εδώ. Υπάρχει η ανάγκη να βρούμε σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ανάγκη παροχής κάποιες επιπλέον στήριξης στους μικρούς παραγωγούς ενώ ταυτόχρονα δεν θα δημιουργήσουμε προβλήματα στη διαρθρωτική προσαρμογή της ε, ευρωπαϊκής ε, γεωργίας. Αυτά είναι τα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και αντικατοπτρίζουν επακριβώς τη νέα προτεραιότητα της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής αλλά και το σύνθετο χαρακτήρα που προκαλεί. Θέλω να επικεντρωθώ και στο θέμα της διακύμανσης των τιμών και της διαχείρισης των αγορών. Η διαχείριση των αγορών είναι ένας όρος ε, πάρα πολύ γενικός που ε, ε, δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα σε όλες τις περιπτώσεις. Η νέα πραγματικότητα είναι οι τιμές των ε, αγροτικών πρώτων υλών είναι ψηλές ιστορικά και θα συνεχίσουν να παραμένουν ψηλές. Άρα όλα τα παραδοσιακά στοιχεία που έχουμε για την παρέμβαση στις αγορές μπορούν να παίξουν το ρόλο μόνο ενός δικτύου ασφαλείας. Ε, ας πούμε, είδαμε τι μπορούμε να κάνουμε με την γαλακτοκομική κρίση. Δεν θέλουμε όμως να παίζουν το ρόλο που έπαιζαν στο παρελθόν και γιατί δεν ε, ε, παρέχουν τα μέσα για να γίνουν ε, οι προσαρμογές που είναι απαραίτητες για τους παραγωγούς. Πρέπει να στοχεύσουμε τα νέα στοιχεία που είναι η μεγαλύτερη τιμή του εισοδήματος και των τιμών. Και εδώ μπαίνουν κάποια δύσκολα ερωτήματα, νέα άγνωστα σε όλους μας, που απαιτούν διαφορετικές απαντήσεις και ενδεχομένως συνδυασμό μέτρων. Στην ανάλυση που θα κάνουμε θα, ε, θα προτείνουμε ε, κάποια πράγματα σχετικά, γιατί για όλα τα κρατημέλη δεν είναι κατάλληλη η διαπάντηση. Κύριε Πρόεδρε, στο σημείο αυτό θα ήθελα να κλείσω θέλω να σας υποσχεθώ ότι στην πορεία της προετοιμασίας της μελέτης επιπτώσεων που θα γίνει βεβαίως πριν την νομοθετική πρόταση θα παράσχουμε οποιασδήποτε ε, επιπλέον πληροφορίες που σχετίζονται με την ανάλυση που θα κάνουμε αλλά και που αφορούν και τη δική σας ανάλυση και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε σε περαιτέρω ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Διευθυντή, τον φίλο μας Τάσο. Ναι, θα πρέπει να εργαστούμε συντονισμένα, όπως και η ομάδα εργασίας που συστάθηκε μαζί με τον Αλβερτές, τον εισηγητή και τους κοιόδης εισηγητές. Όλοι αυτοί θα συνεργαστούν ε, στενή συνεργασία με την Επιτροπή για να επιταχύνουμε την όλη διαδικασία και έτσι η νομοθετική πρόταση της Επιτροπής να μπορέσει να ληφθεί όσο γίνεται, να μπορεί να λάβει υπόψη της όσο γίνεται περισσότερο όλα αυτά τα οποία εμείς ε, ψηφίζουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Έχει ολοκληρωθεί η συζήτηση και δώσαμε τον λόγο στον Τάσο. Και μήπως θα μπορούσε να παραμείνει λίγο ο Άλμπερτ, θα μπορούσε ίσως ο ηγητής να πει ορισμένα πράγματα ακριβώς. Ακούσατε όμως ότι χρειάζεται να αποχωρήσει. Γι' αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε εδώ τη συζήτηση για την αναθεώρηση της ΚΑΠ μετά το 2013 ένα μικρό διαλυματάκι, λίγα λεπτά και μόλις ο Τζορτζ Λάιον θα έλθει εδώ μαζί με τους εμπειρογνώμονες από την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν θα έρθουν εδώ για να εξετάσουμε το επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης ε, για τους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Ευχαριστώ. Σε λίγα λεπτά.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

τροποποίηση της οδηγίας. Ε, παρακαλώ, παρακαλώ στη θέση σας. Ησυχία. Τροποποίηση οδηγίας 2001. Δυνατότητες κρατών μελών να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στην επικράτειά τους. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων μετά από αυτό το λεπτό θέμα που εξετάσαμε το τέλος του Οκτωβρίου, να που μπήκαν στη μέση και καινούρια στοιχεία. Ακούσαμε τις αρνητικές αντιδράσεις των Υπουργών Γεωργίας και Περιβάλλοντος, νομική υπηρεσία του Συμβουλίου που άσκησε δρυμία κριτική κατά των προτάσεων της Επιτροπής. Δύο εκπροσώπους της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου μας έχουμε εδώ. Μαρία Γκόμες Λεάλ και την κυρία Ιωάννα Αναστοπούλου που θα παρουσιάσουν ε, την ανάλυση της δικής μας νομικής υπηρεσίας και μετά θα υποβάλω ορισμένα ερωτήματα μου το ζήτησε ο Τζορς Λάιον που δεν κατάφερε να έρθει εδώ για να ακούσω και τις απόψεις ε, πάνω σε ορισμένα θέματα που ήδη είχε ετοιμάσει ο εισηγητής μας νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου Παρακαλώ, όσο γίνεται πιο σύντομα τα επιχειρήματά σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Λεάλ. ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. μετά από το αίτημα της αρμόδιας επιτροπής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, θα είμαι σύντομη και δεν θα επαναλάβω όλα αυτά που γραπτός έχουμε εξηγήσει. Έχει να κάνει με το αίτημα της Επιτροπής Περιβάλλοντος ότι ανησυχούν σαν για τη νομική βάση της πρότασης αυτής. Η πρόταση αυτή μεταβάλλει την οδηγία 2001-18, τη δυνατότητα ε, των κρατών κλπ. Και ένα εναρμονισμένο σύστημα σχετικά με την ε, κινδύνους για την υγεία και την ε, περιβάλλον και αυτό ώστε τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να απαγορεύσουν στην επικράτειά του σε αυτούς του γενικούς, της γενετικά τροποποιημένου οργανισμούς. Η τυπικότητα τη αγορα και τα προϊόντα τα οποία ανταποκρίνονται σε αυτές τις συνθήκες μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα στην εσωτερική αγορά. Πρόκειται για τυπική ρήτρα εδώ και ανταποκρίνεται στην νομική βάση που έχει με επιλέξει για την εσωτερική αγορά το 114 τη Συνθήκη της Αβώνας. και σύμφωνα με την ομολογία. Η νομική βάση θα πρέπει να συμβαδίζει με το στόχο και το περιεχόμενο και ανταποκρίνεται σε αυτό τις οδηγίες. Προτείνει η Επιτροπή η οδηγία αυτή να αλλάξει με ένα νέο άρθρο στα πλαίσια τα υπάρχοντα και τα ρυθμιστικά πλαίσια ακριβώς. Η πρόταση αυτή τροποποίησης νομίζουμε ότι εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο με τον ίδιο στόχο και δεν αλλάζει ουσιαστικά αυτό το γενικό πλαίσιο. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει ασκής πλευράς και αυτό βάσει της υπάρχουσας νομικής βάσης. Κατά την άποψή μας εξηγήσαμε κάπως τι ακριβώς σημαίνει η νέα αυτή πρόταση της Επιτροπής με το νέο άρθρο που προτείνει την προσθήκη του και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υιοθετήσουν ε, ε, περιοριστικά μέτρα σχετικά με τους γενικά τροπονές που σύμφωνα με την ορισμένη διαδικασία έχουν ε, υιοθετηθεί και χωρίς κινδύνους που να και αυτό σύμφωνα και με τη συνθήκη και θελήσαμε να εξηγήσουμε ότι σύμφωνα με τις συνθήκες σημαίνει σύμφωνα με τις συνθήκες με την νομική του ερμηνεία. Και το άρθρο αυτό που προτείνει τώρα η Επιτροπή είναι περιοριστικά μέτρα στον ε, και στην εσωτερική αγορά θα πρέπει ακριβώς περιοριστικά να ερμηνεύεται και τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να διευθύνουν, να διευρύνουν το νόημά της στην ερμηνεία του αυτού του άρθρου. Και αυτό αν γίνει θα πρέπει να γίνει για επιτακτικούς λόγους ε, γενικού ενδιαφέροντος ε, και όχι έτσι οικονομικούς ε, και αυτό κάθε φορά που το κράτος μάλλον λέει ότι υπάρχει ένας λόγος γενικού ενδιαφέροντος για περιορισμού στην εσωτερική αγορά ε, κάνει μια λεπτομερή ανάλυση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να δει αν ισχύουν αυτά, αν στέκουν. Αλλά γι' αυτό τα μέτρα θα πρέπει να είναι αναλογικό, δηλαδή το περιστικό μέτρο δεν θα πρέπει να προχωράει περισσότερο από το απαιτούμενα για να προστατεύσει τα ε, συμφέροντα αυτά που αναφέρονται και σημαίνει μια εκτίμηση για να δούμε μήπως θα μπορούσε να υπάρξει ένα λιγότερο περιοριστικό μέτρο που θα μπορούσε όμως να ρυθμίσει την κατάσταση. Όταν τα κρατημέλη θα κάνουν χρήση του άρθρου αυτού, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ε, τις ε, προϋποθέσεις ε, που μας, που ζητούνται από την ερμηνεία της συνθήκης. Άρα λοιπόν κύριε Πρόεδρε δεν υπάρχει κανένα νομικό κόλλημα για την νομική βάση. Το μόνο, αλλά εντάξει, είναι τεχνική πολιτική αντιμετώπιση. Να δούμε ακριβώ η ουσιαστική χρήση, η χρησιμότητα, ποια θα ήταν λόγω των περιορισμών που υπάρχουν και ισχύουν στι συνθήκε και όπως έχει τώρα η συνθήκη και η νομική της ερμηνεία. Και ε, η νομική υπηρεσία της Επιτροπής είναι σε καλύτερη θέση για να μας εξηγήσουν με ποιο τρόπο πιστεύουν ότι θα λειτουργήσει αυτό το άρθρο. Και τώρα ακόμα σχετικά με τη σύσταση για την συνύπαρξη, για να δουν αυτά τα μέτρα μπορούν να συνυπάρξουν ακριβώς στα πλαίσια ε, του ΓΚΕΤ ε, και η συνάδελφος Κινάστοπούλου μπορεί να εξηγήσει περαιτέρω. Είμαι στη διάθεσή σας πάντως για τα ενδεχόμενα ερωτήματά σας. No, Ακούστε κάτι η νομική υπηρεσία τη στιγμή που συμφωνεί. Επειδή σίγουρα υπάρχουν ερωτήσεις που χρήζουν απάντησης ε, και αυτά που έχει συντάξει ο εισηγητής. Θα σας ρωτήσω αυτά τα πράγματα και έτσι στα αυτά που θα πείτε μπορείτε να, μπορούν να αποτελούν ήδη απάντηση στις δικές μου ερωτήσεις. Και στη συνέχεια θα ανοίξουμε τη συζήτηση, θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Πρώτο ερώτημα. και εκπρόσωπο τη Επιτροπή ε, από τη Διευσυγεία θα μπορούσε να απαντήσει. Αυτή η πρόταση είναι απαραίτητη βάσει των συστάσεων της Επιτροπής για την συνύπαρξη αυτή με ευρείε δυνατότητε για τα κράτη-μέλη να περιορίσουν την καλλιέργεια παρομοίων γενικά τροποποιημένων οργανισμών σε ορισμένε περιφέρειες, περιοχέ, μέσω του καταλού καθεστώτου του εύκαμπτου στα πλαίσια αυτή τη συνύπαρξη. Και επειδή από την Επιτροπή επανειλημμένα έχει εκφράσει την άποψη ότι θα πρέπει για το 2012 να επανεξετάσει την ομολογία. Μήπω καλύτερα θα ήταν, και αυτό ρωτάει ο συγητή, να μεταβάλουμε το άρθρο 26α και έτσι οι ρυθμίσει για αυτή την ύπαρξη να είναι, να είναι δεσμευτικά για τα κράτη-μέλη και να εργαστούμε προς ε, περισσότερη ευκαμψία, ευληγησία. Δεύτερο ερώτημα. Επειδή αρκετές εθνικές κυβερνήσεις ε, και είναι μια... Ε, είναι έτοιμες αυτές οι χώρες να απορρίψουν αυτή την πρόταση. Αξίζει να συνεχίσουμε την εργασία μας ή μήπως χάνουμε χρόνο και μόνο. Αυτό ρωτάει ο συγητή μα. Τρίτο ερώτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πώς μπορεί να μεταβάλει μία πρόταση από τη στιγμή που οι γνωμοδοτήσει τη νομική υπηρεσία Συμβουλίου, Κοινοβουλίου και Επιτροπή σχετικά με τη νομική βάση του άρθρου 114 τη συνθήκη εμφανίζονται να είναι έντονα τα άρθρα αυτά αντιφατικά. Και ακόμα, για ποιο λόγο η Επιτροπή με το Συμβούλιο δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη για, τις, ε, ε, για την ομάδα εργασία για τους ε, γεννητικά τροπημένους οργανισμούς ότι θα μπορούσαν να περιορίσουν ή να απαγορεύουν την καλλιέργεια στην επικράτειά τους το σαν αρχή με δικαίωμα στην απόφαση το Κοινοβούλιο θα πρέπει να παρακολουθήσει αυτές τις εξελίξεις για να πάρει μια κατάλληλη απόφαση για αυτό το θέμα και το περιθώριο λιγμών για τα κράτη-μέλη φαίνεται καθαρά σχετικά με την οθέτηση περιοριστικών μέτρων για την καλλιέργεια αυτών είναι περισμένο αυτό το πλαίσιο και δεν ξέρουμε καθαρά τι θα ήταν υπέρ αυτών των περιοριστικών μέτρων. Τι θα τα ευνοούσαν. Και ακόμα κάτι απαιτείται περισσότερη σαφήνεια επειδή υπάρχει αυτός, ε, αυτή υπάρχει αντίθεση στην, ε, στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου σχετικά με αυτή την πρόταση. Τι γίνεται, πώς μπορούμε να ε, κάνουμε τα πράγματα ξεκάθαρα. Η Επιτροπή στα κράτη-μέλη θα προσφέρει μια κατεύθυνση όπως ζήτησαν αρκετά κράτη στην πρόσφατη συνάντηση του Συμβουλίου και βάσει ορισμένων στοιχείων, σε ορισμένε δημοσιεύσει και αυτά στον παγκόσμιο εμπορίου, όλα αυτά που, εκφράζονται. Τι γίνεται με, τις, με τους σπόρους γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Ε, πώς δικαιολογούνται όλα αυτά αν δεν υπάρξουν λόγοι πραγματικά επιστημονικοί. Και ακόμα δύο σύντομες ερωτήσεις. Όταν ένα κράτος μέλος ακριβώς θα πρέπει να απαντήσει σε μια διαμαρτυρία που έρχεται από του Ελευθερίου Μπορείου, Μέχρι ποιου σημείου είναι υπεύθυνη η Επιτροπή και θα πρέπει να απαντήσει εκ μέρου μια ε, χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελευταία ερώτηση. Απάντησε η Επιτροπή στη νομική ανακοίνωση του Συμβουλίου. Τι θα γίνει και θα το κάνει αυτό και απέναντι στη νομική υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου. Εντάξει, εμεί εδώ με τη σημερινή μα συνάντηση θα μπορούσαμε να το λύσουμε αυτό. Πρέπει να προσφέρουμε με απάντηση. Αυτέ είναι οι, οι ερωτήσει του George Lyon. Σα τι διάβασα εγώ τι ερωτήσει αυτέ και το λόγο έχει βέβαια και εκπρόσωπος της Επιτροπής. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από την Επιτροπή μάλλον. Και στη συνέχεια μετά η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Η Επιτροπή λοιπόν. Νομική Υπηρεσία επιτροπή. Ο κύριος Πουντέλη. Ναι κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω καταρχήν να πω ότι είμαστε ιδιαίτερως ικανοποιημένοι με την ε, γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου. Κανείς δεν απορεί ότι ε, για το γεγονός ότι με φόβο διαβάσαμε την νομική υπηρεσία, τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου και ε, περιμέναμε ανεπόμονα την νομι, γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Κοινοβουλίου. Όμως αυτή επιβεβαίωσε τη δική μας γνωμοδότηση, τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της Κομισιόν και αυτό μας ικανοποίησε ιδιαίτερα. Τώρα, απαντώντας στο τελευταίο ερώτημα του κ. Ντάιαν, Lion. Δεν ε, θα κάνω επίσημη, θα δώσω επίσημη απάντηση. Δεν ξέρω αν θα ικανοποιήσει η απάντησή μου, αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την άποψη, που, τη γνωμοδότηση που μόλις διάβασε ο εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας, ότι αυτή μας ικανοποιεί πλήρως. Τη σημειώνουμε και δεν έχουμε σκοπό να απαντήσουμε παρά μόνο αν υπάρχει γραπτή επίσημη ε, αίτηση από πλευρά σας. Μπορούμε εδώ να διαβεβαιώσουμε όμως ότι η γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου μας ικανοποιεί. Κατά τα άλλα, το πρώτο ερώτημα. Αν είναι απαραίτητη αυτή η πρόταση. Απαντάμε ναι. Βεβαίως για να ξεκαθαριστεί το νομικό τοπίο, διότι με το παλαιότερο σύστημα αλλά και με το υφιστάμενο σύστημα, αν τα κράτη-μέλη είχαν ε, ρήτρε ε, που αντιέβαιναν ε, την κοινοτική νομοθεσία, προσπαθούσαμε στο επίπεδο Συμβουλίου να αμφισβητήσουμε αυτές τις ε, ρήτρε. Κάθε φορά απέρριπτε απέριπτε αυτές τις νομοθετικές προτάσεις και βρισκόμασταν σε ένα είδος νομικού χάους όπου η Κομισιόν δεν ήθελε να προσφύγει ε, στο δικαστήριο για να καταδικαστούν τα κρατημέλη. Ο πρόεδρος Μπαρόζο ήθελε να βελτιώσει την κατάσταση προτείνοντας ε, αυτό το πακέτο μέτρων στις 13 Ιουλίου, ένα από τα οποία είναι η περίφημη ε, ελευθερία να ε, αποφασίσει ένα κράτος μέλος να πει όχι στην καλλιέργεια στην επικράτειά του. Ε, έχουμε λοιπόν την απόφαση από κάθε κράτος μέλος για να δοθεί έγκριση ή να απαγορευτεί η καλλιέργεια. Χρειάστηκε να διευκρινιστεί η οδηγία και γι' αυτό το λόγο υποβάλαμε την πρόταση ε, τροποποίησης του άρθρου 26β της οδηγίας ώστε το κράτος μέλος να μπορεί να αποφασίζει από μόνο του. Το δεύτερο ερώτημα του κυρίου Λάιονς είναι ποια είναι η ε, μειοψηφία που μπορεί να μπλοκάρει την απόφαση στο Συμβούλιο και αν ε, τίθεται θέμα να χάνουμε ή όχι το χρόνο μας. Δεν μπορώ εγώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Προς το παρόν, στο Συμβούλιο έγιναν ε, στο Συμβούλιο Συζήτησης ε, συζήτηση ε, γεωργίας και περιβάλλοντος. Δεν συμφωνούν πάντα οι απόψεις. Στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη, μια μικρή μειοψηφία που είναι σαφώς αντίθετη. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη ας πούμε περίπου τα μισά που είναι μάλλον υπέρ και τα υπόλοιπα περιμένουν τις απόψεις της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου που είναι μάλλον αρνητική απέναντι στη θέση της Κομισιόν παρά ταύτα ε, ε, ε, όσον αφορά τη νομική βάση. Αλλά όχι μόνο σε σχέση με τη νομική βάση και περιμένουν και την ε, θέση του Κοινοβουλίου. Τώρα, τα κράτη-μέλη έχουν τις τρεις νομικές, ε, τις τρεις απόψεις των νομικών υπηρεσιών, του Συμβουλίου, του Κοινοβουλίου και της Κομισιόν και δεν είμαστε απεσιόδοξοι, εν πάση περιπτώσει, για το αποτέλεσμα. Θεωρούμε ότι δεν χάνουμε το χρόνο μας ε, με το να συζητάμε το θέμα και στη δική σας επιτροπή και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και συνολικά στο Κοινοβούλιο, κύριε Πρόεδρε. Ο Επίτροπος Νταλή επιθυμεί πραγματικά να γίνει συζήτηση επί της ουσίας ε, για την πρόταση αυτή γνωρίζοντας ότι η πρόταση δεν καλύπτει παρά μόνο τις καλλιέργειες και όπως λέει πολύ σωστά η γνωμοδότηση θα γίνει αργότερα μετά από το 2012 συζήτηση για την πλήρη αναθεώρηση της νομοθεσίας για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και δεν θέλουμε τώρα να ξεκινήσουμε αυτή τη συζήτηση για την ε, πλήρη αναθεώρηση ε, της νομοθεσίας. Τώρα θέλουμε να ε, στοχεύσει, να στοχεύσει η συζήτηση το θέμα της καλλιέργειας ή όχι από τα κράτη-μέλη. Τώρα, το άλλο ερώτημα, πώς θα αντιδρά το Κοινοβούλιο όταν, αν είναι αντιφατικές οι τρεις γνωμοδοτήσεις των νομικών υπηρεσιών και πάλι δεν δικό μου θέμα αυτό. Δεν μπορώ να απαντήσω. Τέταρτο ερώτημα. Γιατί δεν συμμερίζεται η Κομισιόν ε, και τους άλλους λόγους που μπορούν να επικαλεστούν τα κράτη-μέλη σε σχέση με την καλλιέργεια αυτή, όπως κάνει το Κοινοβούλιο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πραγματική αντιπαράθεση εδώ. Είμαστε διατεθειμένοι να συμμεριστούμε κι εμείς όπως όλοι. Όπως γνωρίζετε η νομική υπηρεσία κυρίως στηρίζει τις νομοδοτήσεις της θέμα της ε, ε, δημόσιας ε, ηθικής της μογαλιτέ πιμπλίκ υπάρχουν και άλλοι παράγοντες στους οποίους στηριζόμαστε εμείς όπως ας πούμε η διατήρηση των πολιτιστικών ε, και κοινωνικών παραδόσεων η δυνατότητα εξασκήσεως ελέγχου η, ανάγκη ύπαρξης ε, ισορροπίας ε, το γεωργικό χώρο, δηλαδή να υπάρχουν και συμβατικέ καλλιέργειες και βιολογικές καλλιέργειες αλλά και ε, καλλιέργειες γενετικά τροποποιημένων οργανισμών αν το κράτος μέλος ε, επιθυμεί να μην εγκρίνει τι ε, γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες να, και να ευνοήσει τις ε, βιολογικές καλλιέργειες. Όλα αυτά είναι θέματα που πρέπει να μελετηθούν γιατί οπωσδήποτε θα αποτελέσουν αντικείμενο μιας νέας ε, νομολογίας του δικαστηρίου. Δεν μπορούμε να πούμε στα κράτη-μέλη και να τους εγγυηθούμε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε την α ή τη β δικαιολογία. Κανένας δεν θα σας αμφισβητήσει. Εσείς η τεχνική νομική υπηρεσία του της Κομισιόν δεν μπορεί να εγγυηθεί στο κράτη μέλος ότι αν ε, επικαλεστεί τον α ή τον β λόγο πέρα από το δημόσιο αγαθό δεν θα τους ε, αμφισβητήσει κανένας. Αυτό κάθε νομικός θα το καταλάβει. Είμαστε διατεθειμένοι να ε, μοιραστούμε μαζί σας προφανώς ε, τις κατευθύνσεις που θα ακολουθήσουμε σε αυτό το τομέα. Πέμπτο ερώτημα αφορά τη σύγκρουση με, τους, ε, τη σύγκρουση με τον ΠΟΕ. σκεφτόμαστε ότι οι θέσεις και κατόπιν οι αποφάσεις θα πάρουν τα κράτη-μέλη είναι συμβατές με τους κανόνες του ΠΟΕ. Φυσικά και σε αυτή την περίπτωση κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί, ούτε καν εμείς, ότι θα, δεν θα υπάρξει ένα κράτος μέλος του ΠΟΕ, μια τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα αμφισβητήσει, θα προσφύγει κατά ενός ε, ΑΒ κράτους Ευρωπαϊκή Ένωση που θα εγκρίνει κάποιο τέτοιο μέτρο. Τα έξι κράτη-μέλη που έχουν ε, λάβει μέτρα απαγόρευσης ε, της καλλιέργειας του αραβοσίτου Μονσάτο δεν υπέστησαν επίθεση στον ΠΟΕ από τρίτη Τη χώρα, ε, μέλος του ΠΟΕ. Θεωρούμε ότι η δικαιολογία αυτή πρέπει, η δικαιολόγηση πρέπει να εκπονηθεί σωστά, αλλά οπωσδήποτε είναι συμβατή ε, με τα διάφορα άρθρα του κανονισμού του ΠΟΕ και προφανώς απαντώντας στο, ερώτημα 6 αν ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, δεχθεί επίθεση στα πλαίσια του ΠΟΕ από μια τρίτη χώρα για λόγους διακρίσεων κλπ εμείς θα βοηθήσουμε το κράτος μέλος να αμυνθεί θα το βοηθήσουμε. Αυτή τη δέσμευση την έχουμε ήδη αναβάλει. Ο Επίτροπος Ντάλι το είπε εξάλλου δημόσια και θα φροντίσουμε να το βοηθήσουμε ε, να αντιμετωπίσει στεναρά τις ε, επιθέσεις κάποιου τρίτους κράτους, τρίτου κράτους μέλους. Αυτά με δύο λόγια κύριε Πρόεδρε ως απάντηση στα επτά ερωτήματα του κυρίου Λάιον που ε, ε, παρότι λείπει σήμερα, ε, ε, χαιρόμαστε πολύ που μπορέσαμε να τα απαντήσουμε. Ευχαριστώ. Πολύ καλά. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Επιτροπή, την νομική της υπηρεσία για τις απαντήσεις αυτές που μας πρόσφερε. Ξεκινάμε τη συζήτηση. Βέβαια η νομική υπηρεσία όταν θεωρεί απαραίτητο μπορεί να ζητήσει το λόγο. Στεφάν Λεφόλ, πρώτος. Και εγώ λυπάμαι που δεν μπορεί να έρθει λόγω του χιονιού ο George Lyon εδώ. Θα ήθελα να αναγνωρίσω την εργασία του και να το εκφράσω τη φιλία μου. Λοιπόν, μετά από αυτά, τι παραμένει τώρα. Ένα πρόβλημα, το πρόβλημα το οποίο τίθεται. Ακούω την νομική αυτή συζήτηση, είναι υψηλού επίπεδου, υπάρχουν λεπτά λεπτές, ε, ιδιαίτερα λεπτές αναφόρες νομικές στο ύψος ακριβώς και της πολιτικής δυσκολίας. Έτσι, αυτό είναι και το όλο θέμα. Γιατί υπάρχει ένα πολιτικό πρόβλημα πίσω από τα επιχείρηματα τα νομικά, έτσι σχετικά με τους γενικά τροπομένους οργανισμούς. Αυτό δεν αποτελεί μόνο ένα θέμα ρυθμίσεων αλλά και γενική σύλληψης, αντίληψης σχετικά με τη γεωργία, ε, μέσω και της πρόοδου της επιστημονικής. Ε, η δικιά μου άποψη είναι η εξής. Αυτό που μας ρωτάτε είναι γιατί μπορεί να απαγορεύσει ένα κράτος ε, το να χρησιμοποιήσει σπόρους Όπω το είπε και ο πρόσωπο τη Επιτροπή, δεν έχει να κάνει με το σύνολο των γενικά τρομερών οργανισμών, αλλά με του σπόρου και βάσει των όσων μέχρι σήμερα υπάρχουν νομικά αυτό το ναι το όχι σχετικά με αυτό το θέμα εντάξει δεν μπορεί κανείς να έχει αναφορά σε περιβαλλοντικά θέματα ή υγείας αλλά μπορεί να το δικαιολογήσει βάσει διαφορετικών κριτηρίων κοινωνικών, οικονομικών και στρατηγικής επιλογής επίσης σε σχέση με τη βιολογική καλλιέργεια. Αν ισχύει αυτό και αν δικαιολογείται σχετικά με τις επιλογές αυτές. Και γιατί να μην μπορούμε να το βρούμε έτσι και θετικά και σχετικά με, με κάτι θα πρέπει να κάνει κανείς μια επιλογή για να προστατεύσει ή να αναπτύξει την βιολογική καλλιέργεια. Εντάξει, μπορεί να πει όχι στι γενικά τελευταίες οργανισμούς και μπορεί να το αναφέρει αυτό καθαρά, να το γράψει, να το βάλει κάτω γραπτά. Τι γίνεται, αυτό αποτελεί μια σημαντική πρόοδο, τουλάχιστον κατά την απόψή μου. Και στο κάτω-κάτω της γραφής. Στη συζήτηση αυτή δεν πρέπει να είμαστε μόνο στο πλαίσιο μιας άρνησης ε, των γιγαντροπών εργασμών, αλλά να οργανώσουμε τουλάχιστον στην Ευρώπη τη συνύπαρξη. Τι γίνεται σε σχέση με άλλες υπήρους και άλλες χώρες ε, κάνει γεωρικές επιλογές και τελικά ασκεί μια πολιτική ποιοτική μεν η οποία όμως διαβρώνεται ιδιαίτερα από την χρήση γενικά τροπομένων οργανισμών. Ε, αυτό παίζεται, αυτό πρέπει να προστατεύσουμε και μια ρύθμιση γίνεται επειδή είμαστε ικανοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να επιτρέψουμε τη συνύπαρξη και να προστατεύσουμε ότι δεν είναι γενετικά τροπομένος οργανισμός. Α, λοιπόν, ε, το ρωτάω και πάλι. Ναι, το ρωτάω και πάλι. Γιατί. Τι γίνεται, να πούμε καθαρά. Γιατί να αναβάζουμε καθαρά σε αυτά που είναι μέσα. Εντάξει, όταν θέλουμε να έχουμε μια βελεκαλημέρια για μια πολιτική, κοινωνικο-οικονομική προς τη μία κατεύθυνση την άλλη. Γιατί να μην ε, παγορεύουμε τη χρήση αυτών. Και έτσι νομικά νομίζω ότι στέκει περισσότερο, έχει πιο γερές βάσεις. Ο κύριος Άγνιο. Ευχαριστώ. Αυτή είναι μια εξαιρετική κατάσταση όπου η επιστήμη συγκρούεται με το συνέστημα. Κατακέφαλα. Και θέλω να ρωτήσω την νομική υπηρεσία, γιατί ο ΠΟΕ ξαφνικά εμφανίζεται στη συζήτηση. Σίγουρα ο ΠΟΕ θα πρέπει να συνεισφέρει, να εμπλακεί τώρα διότι αυτή τη στιγμή ε, τα βιολογικά τροποποιημένα, τα GMOs, ε, συζητιούνται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες εδώ και πολύ καιρό. Πώς ξαφνικά λοιπόν παρουσιάστηκε ο ΠΟΕ εδώ τώρα που, πρόκειται να αναλυφθούν αποφάσεις. Ε, σκέφτομαι τις, τα επιχειρήματα που είπε η Κομισιόν για τα κράτη-μέλη για να μην καλλιεργούν τα GMO, τα GMOs, συν, πλην, υπέρ, κατά κλπ. Ε, τα επιχείρηματα αυτά δεν είναι συγκεκριμένα. Είναι λίγο μπλεγμένα, λίγο συγκεχημένα. Από την άλλη πλευρά έχουμε το Greenpeace, η οποία στην αρχή ήταν η οργάνωση που τέθηκε επικεφαλής του αγώνα κατά των τροποποιημένων προϊόντων με μεγάλη φασαρία και Είχαμε και εκπροσώπους της Greenpeace που επίσημα δήλωσαν στα μέσα ενημέρωση στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι λάθος τα είχαμε πει τότε και σφάλαμε. Σε μερικά χρόνια λοιπόν θα αναγκαστούμε να πάμε στα δικαστήρια Εν τω μεταξύ η δημόσια αντίσταση κατά των προϊόντων αυτών θα έχει σταματήσει και εμείς θα βρεθούμε μπλεγμένοι στα δικαστήρια λόγω των, ε, του, του μπλεξίματος. Τι είναι λοιπόν καλύτερα, να έχουμε μία βιολογική πατάτα την οποία έχουν, ε, έχει σερίσει οι μύκητες και είναι μαύρη και σάπια ή μία γενετικά τροποποιημένη γη πατάτα. Ε, θέλω να σας απαντήσω ότι υπάρχουν ε, ε, βιολογικά προϊόντα, πατάτες που είτε, είτε τρώγονται είτε δεν τρώγονται. Δεν είμαστε στην παλιά εποχή των βιολογικών. Πρέπει να επανεξετάσετε τα δεδομένα σας. Ε? Η κυρία Μαγκίνας. Ευχαριστώ. Θέλω να, να κάνω μια διατησία μεταξύ των δύο πόψεων. Η παραδοσιακή η γεωργία υπερισχύει. Και ανησυχώ ιδιαίτερα όταν βλέπω αυτή τη συζήτηση να τραβάει στα άκρα και να λέει μία πλευρά ότι εγώ είμαι καλύτερη από την άλλη. Μην ξεχνάτε ε, τον Ιρλανδικό λοιμό, ο οποίος θέρισε ε, χιλιάδες ανθρώπους όταν καταστράφηκε η Σοδιά. Εάν ε, υπάρχει η πιθανότητα να έχουμε βιολογική πατάτα η οποία όμως να μπορεί να παραμείνει υγιής χωρίς να ψεκασμό βεβαίως θα το θέλαμε αυτό πάρα πολύ το θέμα είναι συναισθηματικό αγγίζει του καθενός τα συναισθήματα εμείς χρειαζόμαστε πρωτεΐνες, χρειαζόμαστε σόγια για να ταΐσουμε τα ζώα μας. Άρα λοιπόν ήδη χρησιμοποιούνται τροποποιημένα προϊόντα για την ε, για ε, τροφή των ζώων, για ζωοτροφές. Τώρα και εγώ μπερδευτικά με τα νομικά επιχειρήματα, αλλά αναρωτιέμαι μήπως η συζήτηση αυτή είναι πρόορη, δεδομένου ότι και το Συμβούλιο αυτή τη στιγμή μελετά την κατεύθυνση της πρότασης. Αν και καταλαβαίνω γιατί η Κομισιόν παρακινήθηκε να υποβάλει μια πρόταση σε αυτό το θέμα. Υπάρχει πρόβλημα, όντως, για κράτη-μέλη τα οποία δεν θέλουν να καλλιεργήσουν τροποποιημένα. Για άλλα κράτη το θέμα δεν έχει υπάρξει, δεν έχει δημιουργηθεί το θέμα της συνύπαρξης ε, στην, ε, στον αγροτικό τομέα νομίζω μπορεί να χρησιμοποιηθεί το επιχείρημα της συνύπαρξης. Αλλά πριν γίνει αυτό πρέπει να έχουμε καλύτερη ενημέρωση. Καλύτερη ενημέρωση και πληροφόρηση των παραγωγών μας και πρέπει να ξεπεράσουμε και νομικά εμπόδια. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα στην εσωτερική αγορά. Εάν αφήσουμε τα κράτη-μέλη να διαλέξουν τα σημεία που τους αρέσουν και να διαγράψουν τα άλλα, θα δημιουργήσουμε ανισότητες στην αγορά. Και μέσα στην, στις μεταρρυθμίσεις της ΚΑΠ, όπου ζητούμε περισσότερη ευελιξία για τα κράτη-μέλη, και αυτό το στοιχείο της ευελιξίας δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Να υπάρξει λοιπόν, να υπάρχει αυτό το στοιχείο. Μία σύντομη παρατήρηση. Όταν ακούω ότι υπάρχουν και κοινωνικό κοινωνικά κριτήρια μέσα σε ένα οικονομικό πλαίσιο παθαίνω πονάει το στομάχι μου. Ε, διότι η κοινωνία αλλάζει απόψεις, έτσι. Λοιπόν, όταν θέλουμε να εφαρμόσουμε κοινωνικά πολιτιστικά κριτήρια, η κοινή γνώμη σήμερα είναι θετική, αύριο είναι αρνητική και τα Λοιπόν, εγώ πιστεύω εάν ε, νομικά επιχειρήματα εμπλέξουν κοινωνικοπολιτιστικές πτυχές, ε, δεν θα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, οπότε δίνω και πάλι το λόγο στην Κομισιόν να απαντήσει στα ερωτήματα που τέθηκαν. Ευχαριστώ. Ναι κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ακούσαμε διάφορες ερωτήσεις και αρκετά σχόλια για τις ερωτήσεις του κύριου Λεφόλ. Ο πρόεδρος Μπαρόζο το Σεπτέμβριο του 2009 στο πρόγραμμα που παρουσίασε για την επανεκλογή του μίλησε καθαρά για αυτές τις ελεύθερες καλλιέργειες. Τι σημαίνει αυτό. Ναι, για τα κράτη-μέλη που δεν επιθυμούν να καλλιεργήσουν και όχι το αντίθετο. Δεν είναι εκείνοι που θέλουν να καλλιεργήσουν που θα πρέπει να κάνουν ειδική αίτηση. Μετά από την έρευνα από την ΕΦΣΑ, από το επιστημονικό όργανο δηλαδή για τους γενικά τροποποιημένους οργανισμούς που αποδείχτηκε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από αυτούς, ας πούμε, επανασχάρη για την υγεία των ζώων, των ανθρώπων, του περιβάλλοντος. Τι μας λέει η επιστήμη. Ότι ο γενικά τροποποιημένος οργανισμός είναι υγιής και σίγουρος. Δεν υπάρχει πρόβλημα κίνδυνος. Και σαν επιλογή στρατηγική ποια ήταν εκείνη που δεν επιθυμούν να προχωρήσουν στην καλλιέργεια να πάρουν μια νομική φύσεως απόφαση σε εθνικό επίπεδο ή σε περιφερειακό επίπεδο. Γιατί και μια περιφέρεια ενός κράτους μέλους μπορεί να λάβει παρόμοια απόφαση και να καλύψει αυτή η απαγόρευση μόνο αυτή την περιφέρεια και όχι το σύνολο του κράτους μέλους της επικρατείας του. Αυτή η επιλογή στρατηγική λοιπόν έγινε και έτσι αποδεικνύεται ότι τον πρώτο λόγο στην υπόθεση την έχει, τον έχει επιστήμη θα πρέπει να ξεκαθαρίζει ότι ο γενετικός τροπημένος οργανισμός είναι ασφαλής. Αν υπάρχει ένα κίνδυνος, επαναλαμβάνω, για τα φυτά, τα ζώα, τον άνθρωπο κλπ. Αν υπάρχει ένα κίνδυνος, σίγουρα τότε δεν θα επιτραπεί. Για τους σπόρους τώρα. Η απαγόρευση της ελεύθερης κυκλοφορίας σπόρων δεν θίγεται αυτή, αλλά η σπορά οι γενικά τροπομένοι σπόροι μπορούν να κυκλοφορούν ε, έστω και σε μια περιοχή, σε ένα κράτος μέλος που απαγορεύει τη φύτευση, τη, τη, την καλλιέργεια, τη σπορά. Και έτσι εξηγείται και η στρατηγική αυτή η νέα. Αρμοδιότητα βέβαια των κρατών μελών είναι να αιτιολογήσουν τη σχετική απαγόρευση λέτε γιατί να, μην είμαστε, γιατί να είμαστε πιο ξεκάθαροι. Ναι, στο δεύτερο έγγραφο μαζί αυτό εδώ, 13 Ιουλίου, όλα αυτά που δόθηκαν για τη συνύπαρξη, ας την πούμε έτσι, σε εισαγωγικά. Τον όρο τον αλλάξαμε του πρώτου εγγράφου για αυτή την ε, συνύπαρξη. Ήταν κάπως περιορισμένο. Η διαφορά ανάμεσα σε σπορά, ανάμεσα στην αγρο βιολογική καλλιέργεια, στους γενικούς οργανισμούς κτλ. Είχε το κατάλληλο πλαίσιο και προσφέραμε περισσότερη ελευθερία στα κράτη-μέλη ώστε να χαράξουν τους κανόνες ε, σποράς ανάμεσα στις δύο αυτό και να είναι πολύ ευρύτερο το πλαίσιο Ιδιαίτερε δυνατότητες χρησιμοποίηση αυτού του κειμένου ώστε να υπάρξει αυτή η διαφοροποίηση. Το ίδιο ισχύει και για το κατόφλι μόλυνσης. Ρώτησε γιατί αυτά μπαίνουν στα πλαίσια της συζήτησης. Εάν υπάρξει μια παγόρευση μιας καλλιέργειας που δεν βασίζεται επιστημονικά, υπεύθυνοι του Διεθνούς Εμπορίου και σε εμά επίσης στη Γενική διεθνή Εμπορίου ε, εξέφραν την ασυχία τους γιατί Μήπως αυτές οι απαγορεύσεις θέσουν σε κίνδυνο τη σχετική ισορροπία με τους εταίρους μας, τους εμπορικούς και να υπάρξουν ε, και ε, προσφυγές και κατηγορίες ε, στον ΠΟΕ που δυσκολεύουν και τη θέση των κατωμελών και της, και, του, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είδαμε για τις ορμόνες και από τη στιγμή που αποφασίστηκε η διατήρηση αυτής της απαγόρευσης να χρησιμοποιούνται οι ορμόνες οι αυξητικές ζώα. Από την άλλη μεριά, αντισταθμητικά ποσά και μάλιστα υψηλά στι ΗΠΑ που χρειάζεται να πληρώσει. Άρα λοιπόν όλα αυτά επηρεάζουν την κατάσταση στον ΠΟΕ και στο διεθνέ εμπόριο. Είναι σημαντικά λοιπόν και να αποφύγουμε τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο να μπουν σε ένα δρόμο και να έχουμε τελικά οικονομικά προβλήματα απέναντι στι τρίτε χώρε. Έτσι σε γενικές γραμμές και σύντομα σύντομα νομίζω ότι απάντησα κύριε Πρόεδρε στις ερωτήσει σας. Ευχαριστώ την Κομισιόν. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων. Η επόμενη μας συνεδρίαση θα είναι στις 25 Ιανουαρίου 2011 στις 3 και 26 Ιανουαρίου όλη τη μέρα. 9 η πρωινή και 3 η ώρα η απογευματινή.